Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Αλληλία της Νέας Θητείας. Ελπίζω να περάσατε όλοι καλό καλοκαίρι και να θέλετε πολύ να ψηφίσετε. Ένας ε, συνάδελφος ε, νέος είπε «Μα ψήφισα 40 φορές σε μια επιτροπή, ποτέ δεν έχω ψηφίσει 40 φορές». Ε, εγώ όμως που είμαι παλιός, εδώ και 15 χρόνια Έχω δει προέδρου να τα πηγαίνουν χάλια στις ε, ψηφοφορίες και τώρα να δω πώς θα τα πάω εγώ. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε το πρώτο θέμα τη ημερήσιας διάταξη. που είναι ακριβώ η έγκριση τη ημερήσιας διάταξη. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, προτείνω να την εγκρίνουμε. Εγκρίνεται, ευχαριστώ πολύ. Και το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών της 23ης Ιουλίου τρέχοντος. Αν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνονται και τα πρακτικά. Δεν έχω ανακοινώσει ως πρόεδρος. Οπότε περνάμε στις ψηφοφορίες για το γενικό προπολογισμό. Θα χρειαστείτε τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Ελπίζω να τι έχετε όλοι. Καταπληκτικό αν τις έχετε όλοι. Γιατί θα στοιχημάτιζα ότι τουλάχιστον ένας θα την είχε ξεχάσει. Και φοβόμουν πως θα ήμουν εγώ βέβαια. Οπότε, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Έχασα το στοίχημα που θα μπορούσα να έχω βάλει. Λοιπόν, στην ε, τελευταία μας συνεδρίαση 23 Ιουλίου σας παρουσίασα το σχέδιο γνωμοδότησης για το σχέδιο προπολογισμού που πρέπει να αποσταλεί στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ανέλαβα αυτό το ρόλο ως πρόεδρος. Είναι τυπικό. Η γνωμοδότηση αυτή είχε και τις πολιτικές μας προτεραιότητες και τις τροπολογίες μας επί των κονδυλίων του προπολογισμού που μας αφορούν. Χρειάστηκε να υποβάλουμε τροπολογίες μέχρι τις 25 Ιουλίου και για τα δύο τμήματα. Υποβλήθηκαν 62 τροπολογίες στη γνωμοδότηση και 14 για τα κονδύλια του προπολογισμού. Και τώρα θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε τις τροπολογίες επί του προπολογισμού, του γενικού προπολογισμού. Πρώτο θέμα είναι το 11.03.01 για τη γραμμή του προπολογισμού 11.03.01 άρχεται η ψηφοφορία. Να σας δώσω χρόνο γιατί είναι η πρώτη μας ψηφοφορία. Εντάξει. Ωραία, ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Το επόμενο είναι το 11.01.02.01. Άρχεται. Πέρασε. τις προφορίες. Εγκρίνεται. Το επόμενο. 11.01.01. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 11.01.03. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 11.06.62.01 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 11.06.64 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 11-06-63-01 άρχεται πέρας απορρίπτεται 11-06-77-18 άρχεται πέρας δεκτή 11.06 77 19 άρχεται πέρας δεκτή 11.06 77 21 άρχεται πέρας απορρίπτεται 11.06 77 22 άρχεται Πέρασε. Δεκτή. 11.06, 77, 23. Άρχεται. περασε Απορρίπτεται. 11.06, 77, 24. Άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. 11-06-77-20 77 20 άρχεται περασε δεκτή ευχαριστώ πολύ συναρπαστικό ε? όχι ωραία Οπότε, οπότε, τροπολογίες επί της γνωμοδοτήσεως. Τονίζω ότι όπως είπε ο κ. Κόρμπετ και επιβιώνει η γραμματεία, η τροπολογία 57 είναι συμβατή με τις 53 και 55 και 54. Θα γίνει μια διόρθωση στο κατάλογο ψηφοφοριών αν χρειαστεί. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στην τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρασε. Α, ναι, λίγο περισσότερο χρόνο θέλετε. Ωραία, άρχεται. Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία. Κυρία Κιλέρα, έχετε έναν παραπάνω που ψηφίζει. Μπορείτε να δείτε Ποιοι ψηφίζουν με τους σοσιαλιστές. Εντάξει. Μάλιστα. «25 ψήφισαν, καταπίπτει. Απορρίπτεται δηλαδή. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ε, ψηφίζουμε. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Α, με συγχωρείτε. Πάμε στην 10 ψηφίζουμε. Πέρας. Πέρας ψηφοφορίες απορρίπτεται. Τι γίνεται τώρα. Τροπολογία 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Τροπολογία 13. 16. 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ψηφίζουμε. Πέρας. Τροπολογία 17. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Ε, ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκαν λοιπόν με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, 27. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. 28. Ε, ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 32. Τροπολογία 32. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην προφορική τροπολογία. Κόντε Ταρδίνο. Έχετε την προφορική αυτή γραπτή στο κατάλογο ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιο νούμερο ήταν, παράγραφος 6α, προφορική τροπολογία και θα πρέπει να είναι στον κατάλογο ψηφοφορία σας. Εντάξει κυρία Κιλέρα, μάλιστα. Ωραία λοιπόν, ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Βίκυ, 36. Ε, vote is open. Vote is closed. Εγκρίνεται. Η 37 τώρα είναι μια προσθήκη. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 43. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 42. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 44. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 45. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. 47. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 48. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. 53 Έκρινεται. Πάμε τώρα στη 57. Κόρμπετ. 57 Κόρμπετ ψηφίζουμε. Ναι, κύριε Μιγιάν μόνο. 57 ψηφίζουμε. Ε, Πέρασε τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 58 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 59 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60 ε, ε, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 61. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Τροπολογία 62. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 25 ψήφοι υπέρ, 0 κατά, μία αποχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα μπορείτε να βάλετε στη θέση τους τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Now, where, where's the commission? Uh, Στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο 6 της ημερήσιας ε, ε, διάταξης που αφορά τα θέματα της αλίας, ε, της μονομερής αλίευσης κουμπρίου από την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Οι κυβερνήσεις των δύο αυτών χωρών ανήγγειλαν τον Ιούνιο ότι θα αυξήσουν το ποσοστό αλλιεύματος σκουμπριού. Αύξησαν λοιπόν την ποσόστοση που είχαν, πράγμα το οποίο επηρεάζει την βιωσιμότητα και την ε, κέρδη τα οποία μπορούν να έχουν οι δικοί μας ε, αλείς. Έχουμε τον, μαζί μας τον κύριο Φαμπρίτσιο Ντονατέλα, ο οποίος είναι κύριο σύμβουλος της ε, συμφωνίας για τις αλίες της βόρειας χώρες από την DG Mare και Εδώ και πέντε χρόνια αυτό συζητούμε το θέμα και πριν από πέντε χρόνια. Ίσως ήταν πολύ μικρότερες οι ποσότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει ο πόλεμος για το σκουμπρί. Κύριε Ντονατέλα, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που μας επιτρέπει να δώσουμε πληροφορίες στην Επιτροπή σας για το τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά το σκουμπρί και τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία, η Γρυλανδία, η Νύση, η Φέροε και η Ισλανδία αλλιεύουν. Και να σας πω ποιες είναι οι συζητήσεις που έχουμε με τις διάφορες παράκτιες χώρες για τα αποθέματα σκουμπριού. Στο παρελθόν, για το σκουμπρί υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις και όπως θα θυμάστε και πρόσφατα, λύθησαν διάφορες πρωτοβουλίες από κάποιες χώρες δεδομένου ότι υπήρχαν κάποιες ε, αυξήσεις των ποσοστώσεων που ελήφθησαν μονομερώς από κάποιες από αυτές τις χώρες. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αναφέρω είναι ότι το σκουμπρί είναι θέμα συζητήσεων και διαγραπανωτέσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω τα πρόσφατα γεγονότα διότι έτσι θα καταλάβετε ίσως καλύτερα την κατάσταση. Το 2014 υπήρξαν εκτενείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφόρων παρακτήων χωρών, δηλαδή των χωρών που έχουν το δικαίωμα να αλλιεύουν τα ψάρια αυτά και συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις χώρες την Ισλανδία και αργότερα την Γρυλανδία που προσφάσισαν να συμφωνήσουν για το πώς θα κατανείμουν τα αποθέματα βάσει ποιου συστήματος ποσοστώσεων, αν κάνουμε κάποια σύγκριση, θα μπορούσα να πω ότι προσπαθούν να επιτύχουν γι' αυτό το πελαγικό είδος μία κάποια σταθερότητα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και δύσκολα τελικά κατέληξαν σε συμφωνία. Μόνο η Νορβηγία και η Νύση Φεροέ συμφώνησαν και άφησαν ένα παραθυράκι ανοιχτό στις άλλες χώρες για να μπορέσουν η Γρυλανδία και η Ρωσία να μπορέσουν να συμφωνήσουν. Οι χώρες αυτές ε, ε, βεβαίως αλλιεύουν σε εκτός των χωρικών τους υδάτους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλησαν για αυτές τις άλλες παράκτητες χώρες, όπως σας είπα, οι δύο πρώτες χώρες να αφήσουν ένα παραθυράκι ανοιχτό. Αυτό, λοιπόν, είναι, αυτή είναι η κατάσταση το 2014. Το 2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία και ως το 22 θα παρατεθεί και μπορεί να υπάρξει και ένα συμπληρωματικό έτος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι έτσι μπορεί κανείς να καταλάβει τη σταθερότητα την οποία προσπαθούμε να έχουμε ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα αποθέματα σύμφωνα με τους στόχους περί διασφάλισης των αποθεμάτων και σύμφωνα με αυτά τα οποία μας λένε οι επιστήμονες που γνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, κάποιες χώρες από αυτές δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν, να καταλήξουν. Οι αξιώσει τους όμως δεν ήταν απόλυτα σαφείς και μέχρι πολύ πρόσφατα δεν ήταν καθόλου σαφείς μάλιστα και δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν με μας. Άρα δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν μέρος της συμφωνίας. Και οι ποσοστώσει τους ορίστησαν μονομερός, ήταν σταθερά μέχρι πέρσι. Κάθε χρόνο από το 2014 και μετά η Ισλανδία αποφάσιζε ποια θα ήταν ετησίως, ε, ποιες θα ήταν ετησίως οι ποσοστός και πρέπει να πω ότι αποφάσισε και αυξήσεις από το 14 λοιπόν έως το 19 τουλάχιστον το πρώτο μέρος του έτους 19 πρέπει να πω ότι υπήρχε μία σταθερότητα με την, ε, στον τρόπο με την οποία όριζε η Ισλανδία τις ποσοστώσεις. Αυτά τα πράγματα άλλαξαν όμως τελευταία. Όταν αποφάσισαν οι νήσοι Φεροέ να μην αλλάξουν το ΤΑΚ, πήρε διαφορετική εντελώς άποψη η Ισλανδία. Αντίθετα με αυτά τα οποία είχαμε εμείς αποφασίσει και πρέπει να πω ότι για μας αυτό ήταν αποτέλεσμα σταθερότητα στην αγορά για το 2019 αλλά τώρα βλέπουμε ότι στο 19 ενώ είχαμε αποφασίσει να μην αλλάξουμε τα τάκ, αποφάσισε τις ποσοστώσεις της να τις αυξήσει μονομερός η Ισλανδία σε ποσοστό 21,5% του ΤΑΚ με εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Δεν θέλω εδώ να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι για κάποια χρόνια η Ισλανδία, παρά το γεγονός ότι ήταν μέρος της συμφωνίας, όπως οι άλλες, λάμβανε υπόψη τις αποφάσεις των άλλων χωρών για πρώτη φορά εφέτος αποφάσισε μονομερός να αυξήσει τις ποσεστώσεις, ακολούθησε μια διαφορετική γραμμή και τώρα ποια είναι η κατάσταση παρά το γεγονός ότι η αύξηση του ΤΑΚ είναι 21,5% η αύξηση αυτή δεν βασίζεται σε επιστημονικά ευρήματα. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική με τη Γρυλανδία. Πρώτα απ' όλα <clears throat> διότι ο όγκος της αύξησης δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά στην περίπτωση αυτή η Γρυλανδία σέβεται τα τάκτα που έχουν συμφωνηθεί από τις άλλες χώρες. Παρά το γεγονός ότι αυτό το... αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, η Γρυλανδία επίσης μας εξέπληξε με αυτή την άκρηση και τελευταίο, όχι λιγότερο σημαντικό, έχουμε και μία παρεμφερή απόφαση η οποία ε, λαμβάνεται από τη Ρωσία, που είναι χώρα που αλλιεύει, δεν είναι παράκτια χώρα σαν τις άλλες, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό που συνέβη τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Τρεις χώρες αποφάσισαν να αυξήσουν μονομερός για το σκουμπρί την ποσόστοση αλίευσης Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει αστάθεια στον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων και ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι θα δημιουργηθεί μια κατάσταση σήμερα την οποία οι προσπάθειες που κάνουμε για να διασφαλίσουμε τα αποθέματα τίθενται εν κινδύνο. Με δύο λόγια, η υπεραλίευση ξεπερνάει σε ποσοστό το 25%. Και αυτό είναι το στοιχείο το οποίο θα ήθελα με απόλυτη σαφήνεια να σας εξηγήσω. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία απόφαση που μας κατέλαβε εξαπίνης που είναι αντίθετη με αυτή που πήραν οι τρεις άλλες παράκτιες χώρες για να μπορέσουμε να έχουμε σταθερότητα και τρίτο στοιχείο αυτή τη στιγμή βλέπουμε αύξηση των ποσοστώσεων που πραγματικά θα οδηγήσει σε υπεραλίευση. Συγκεκριμένα του σκουπιού. Κύριε Σκορμπιού. Σκουμπριού. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε μπορώ εδώ να σταματήσω και να αρχίσουμε συζήτηση. Ή θέλετε να σας δώσω και συμπληρωματικά στοιχεία. Ό,τι πιστεύετε εσείς. Ίσως θα ήθελε να ακούσει και την Επιτροπή η Ποια είναι η... εσείς ως Επιτροπή, τι αποφασίζετε να κάνετε. Τώρα, με τις αντιπροσωπείες μας στις χώρες αυτές, στις χώρες αυτές ήρθαμε σε επαφή, ώστε να κάνουμε επίσημα ένα διάβημα κατά της απόφασης αυτής και να διαμαρτυρηθούμε στην Ισλανδία. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε με τη Ρωσία, δεδομένου ότι εδώ δεν μιλούμε με παράκτια χώρα. Το πρώτο στοιχείο ήταν μια πολύ έντονη αντίδραση των δύο παρακτήαχρων από τις τρεις οι δύο συλλογικά αποφάσισαν να στείλουν μια ισχυρή διαμαρτυρία και στη Γρυλανδία και στην Ισλανδία. Ίσως σας φαίνεται γραφειοκρατικό, αλλά μιλούμε για ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ένα πλαίσιο ή μια οργάνωση υπό την οποία εργαζόμεθα. Πρόκειται λοιπόν για ένα συλλογικό μήνυμα που έστειλαν αυτές οι τρεις παράκτιες χώρες ώστε να τους καταστήσουμε σαφές ότι είναι απαράδεκτη αυτή η απόφαση. Δεύτερον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κυρίω Επιτροπή, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, στα πλαίσια της κοινή πολιτικής και σταθερά από νομική βάση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μονομερός. Δηλαδή, ελπίζουμε ότι σε συνεργασία με τις άλλες παράκτιες χώρες και σε συντονισμό θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε επίσης ποιες δράσεις, ποιες ενέργειες μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των αποφάσεων αυτών. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν και τα, κάποια μέλη της Επιτροπής γνωρίζουν είναι ότι το 2013 χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν, και εδώ πολύ προσεκτικά αναφέρω αυτό που λέω, μια κατάσταση η οποία φαίνεται επί χάρτου πάρα πολύ παρεμφερής, αλλά στην πράξη είναι πολύ διαφορετική με τις νήσες Φερόε. Σήμερα λοιπόν προσπαθούμε να μελετήσουμε όλα αυτά τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουμε, ώστε να είναι η ενέργεια που θα αναλάβουμε πολύ πιο δυναμική από άλλες. Πρώτα απ' όλα, Πρώτο βήμα. Δίαυλοι επικοινωνίες με τις χώρες αυτές δεν θα πρέπει να κλείσουν. Στο... Για τον Οκτώβριο θα συζητηθούν και θα καθοριστούν τα τάκ για του χρόνου και είναι προσκεκλημένες όλες οι χώρες για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να δούμε πώς θα το δείσουμε. Σήμερα λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν τεχνικά αλλά και νομικής φύσεως θέματα, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ πλόκο θέμα. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στα πλαίσια των συμφωνιών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα γίνει με τη Γρυλανδία, πώς θα λάβουμε μέτρα. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα επιβάλλουμε κυρώσει, αλλά νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με αυτό τον συγκεκριμένο την το συγκεκριμένο εταίρο, με μια συμπεριφορά η οποία πραγματικά ε, είναι απαράδεκτη. Η ερώτησή μου, όταν λέτε στην Επιτροπή τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας, εννοείται κυρώσεις. Δεύτερον, τι ε, γίνεται με τέτοιου είδου με τη Γρυλανδία και την Ισλανδία. Όταν δούμε ποιες ε, δράσεις, ποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μας, κυρίως αναφέρομαι σε έναν κανονισμό και τελικά στο τέλος της διαδικασίας μπορεί να οδηγηθούμε σε κυρώσεις. Αλλά αν θέλετε θα είναι το ίστατο βήμα που θα λάβουμε. Εάν αποτύχουμε στο μεταξύ διάστημα να βρούμε πρακτικές λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Αντί λοιπόν να εξετάζουμε μια κατάσταση στην οποία ευθύς εξ αρχής θα επιβληθούν κυρώσεις, η οπτική μας είναι να δούμε αν υπάρχουν άλλες δυνατότητες επίλυσης αυτής της διαφοράς. Εάν τελικά δεν γίνει τίποτα, θα επιβληθούν κυρώσεις. Δεύτερον, η συμφωνία με την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε με την Ισλανδία μία συμφωνία στο παρελθόν ότι είναι κάπως λανθάνουσα ε, αυτή η συμφωνία. Πρέπει να πω ότι μέχρι το 2009 ίσως δεν υπήρχε ε, κανένα ενδιαφέρον να ε, μπορέσει αυτή η συμφωνία να ανανεωθεί. Πρόκειται για μια απλού τύπου συμφωνία, αλλά οι δύο εταίροι το 2009 συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνεχιστεί αυτή η συμφωνία. Αυτή λοιπόν τη στιγμή υπάρχει, αλλά είναι σε λανθάνουσα φάση αν θέλετε. Και όσον αφορά την Γρυλανδία, πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε ότι όντως έχουμε μία ε, συνεργασία βιώσιμη αλληλεία είναι διαφορετική από αυτή την οποία έχουμε στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουμε με τις υπόλοιπε παράκτιες χώρε. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη συμφωνία τρόπου ε, κάποιων ε, αλλιευμάτων που δεν είναι απαραίτητο μέλος των πελαγικών ειδών, αλλά δεν αφορούν όλο ιδιαίτερα στο σκουμπρί που πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικά. Και για να ολοκληρώσω, για να μπορέσουμε να κάνουμε διαχείριση των ε, αποθεμάτων σκουμπριού στην Ειδική Επιτροπή ΝΕΡ δεν θέλει για την διαχείριση του σκουμπριού να κάνει τίποτε. Πρόκειται για μια, ένα φόρουμ, μια πλατφόρμα στην οποία συνεχίζονται οι συζητήσεις, αλλά δεν πρόκειται για οργάνωση η οποία ε, μπορεί να λάβει δράση για τέτοιου είδου θέματα που αφορούν τα αποθέματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά σε επίπεδο ε, αυτής της πλατφόρμας μπορούμε να συνεργαστούμε αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην σταματήσουμε τη συνεργασία με αυτός τους εταίρους. Ευχαριστώ. Uh, Καλέσαμε και τον πρέσβη της Ισλανδίας να στείλει εκπρόσωπο. Αλλά η Ισλανδική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να συμμετάσχει. Αλλά απέστειλε ένα σημείο μας όλα τα μέλη μας που παρουσιάζει τη θέση τους και τους είδα κατηδίαν ε, εγώ και θα σε ενημερώσω για όσα διεμήφθησαν. Ωστόσο, καλέσαμε και εκπροσώπους από την Γρυλανδία και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κλάιστ από την μόνιμη αντιπροσωπεία για την ε, παρουσία του. Κύριε Κλάιστ, να σε εξηγήσω το πλαίσιο. Ξέρω ότι αρχές Ιουλίου έμαθε η Επιτροπή ότι η Γρυλανδία αποφάσισε να αυξήσει από 59.000 σε 70.000 την μονομερή ποσόστοσή της για το σκουμπρί, αύξηση δηλαδή 18% που είναι τώρα 11%, 11 περίπου της ε, συνολικής δυνατότητας αλίευσης. Και αυτό ήταν κεραυνός εν εθρία. Η Επιτροπή μας βέβαια πολύ θα ήθελε να ακούσει ε, πώς παρουσιάζεται το θέμα, τα επιχειρήματά σας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αλίας που μας προσκαλέσατε σε αυτή τη συνάντηση για το θέμα ημερησία διάταξη για το σκουμπρί. Είναι προτεραιότητα της Γρυλανδίας να είναι υπεύθυνη και ενεργή ως ε, παράκτιο κράτος. Αυτό αποδεικνύεται από την συνεχή συμμετοχή μας στις διαβουλεύσεις των παρακτήων κρατών ιδιαίτερα για το σκουμπρί. Πιστεύουμε ότι οι διαβουλεύσει και η συνεργασία μεταξύ των ε, παρακτιοκρατών για τα πελαγικά είδη είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για βιώσιμη αλίευση με βάση τα επιστημονικά και αντικειμενικά στοιχεία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό η μονομερής αύξηση των ποσοστώσεων από την Γρυλανδία και την Ισλανδία είναι παραπλανητικός ως τίτλος. Δεν αντανακλά την ενεργό συμμετοχή μας στις διαβουλεύσεις. Πιο αντικειμενική ε, διατύπωση, κατά τη γνώμη μας, θα ήταν καλύτερη. Θα ήταν πιο επικοδομητική και κατάλληλη. Παρ' όλα αυτά, σημειώνουμε ότι εμείς, η Γρυλανδία, όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί για διάλογο για κάθε θέμα και ευχαριστούμε την Προεδρία που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την ε, άποψή μας για το θέμα αυτό. Η Γρυλανδία έγινε αναγνωρισμένο παράκτιο κράτος που συμμετέχει στην Συμφωνία για το Σκουμπρί το φθινόπωρο του 2016. Αλλά ως παρατηρητές συμμετείχαμε στις διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό ήδη από το 2014. Ως παρατηρητές όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία και τα νησιά Φαρόε κατέληξαν σε μία συμφωνία για την αλίευση του σκομπρίου για την περίοδο 14 έως και το 18. Τον, ε, το φθινόπωρο του 18 τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να παραταθεί αυτή η συμφωνία του 2014. Αυτό έγινε χωρίς τη συμμετοχή της Γρυλανδίας και ούτε καν της Ισλανδίας στην συμφωνία για το σκουμπρί από την ε, άποψή μας. Αυτό ήταν μια ευκαιρία που χάθηκε για να υπάρξει μια συμφωνία χωρίς εξαιρέσεις. Η Γρυλανδία λοιπόν δεν έχει υπογράψει. Δεν είναι συμμετέχον κράτος τη συμφωνίας αυτής και ως παράκτιο κράτος έχει δικαίωμα να αποφασίσει την ποσόστοσή της. Τον, ε, στις 5 Ιουλίου η Γρυλανδία αποφάσισε να αυξήσει την ποσόστοση για το 2019 από 59.729 τόνους σε 70.411 τόνους. Ο λόγος για την απόφαση ήταν αναθεωρημένες επιστημονικές σύμβουλες από τον οργανισμό ISIS για το σκουμπρί, για το 19 που από 300.000 318 ε, πήγε στις 370.000 ε, τόνους. Η Ιρλανδία προσάρμοσε την ποσόστοσή της με βάση τα αυξημένα στοιχεία που είχαμε και που συγκεκριμένα έλεγαν ότι είναι 770.358 τόνοι. Όμως είναι προτεραιότητα πάντα της Ιρλανδίας να συμμετέχει στην εργασία για να υπάρξει μια επίσημη συμφωνία για το σκουμπρί με τη συμμετοχή όλων των παρακτήων κρατών, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε μακροχρόνια βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ε, σκουμπριού. Η Γρυλανδία έχει μακροχρόνια συνεργασία με την Ένωση και πιστεύουμε προς είναι προς το συμφέρον όλων μας να διατηρήσουμε καρποφόρα και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο μερών όπως έχουμε και για τις διαβουλεύσεις για άλλα είδη και γενικότερα στους οργανισμούς, ε, τους περιφερειακούς οργανισμούς για την αλληλεία σε αυτή την περιφέρεια. Σε ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σας παρουσιάσω την άποψή μας. Επαναλαμβάνω ότι η Γρυλανδία είναι πάντα ανοιχτή για επικοδομητικό διάλογο για βιώσιμη αλίευση του σκουμπριού. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Ο κύριος Μιγιάν Μόν, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπο της Γρυλανδίας που είχε την ευγένεια να έρθει εδώ να μας ενημερώσει για τη θέση τη, για τη θέση της, ε, των εδαφών που εκπροσωπεί εγώ. Ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη λύπη μου για αυτές τις μονομερείς αποφάσεις αυτών των δύο ε, συμμετεχόντων να αυξήσουν ε, την ποσόστοσή τους. Εάν θέλουμε να είμαστε υπέρ της βιώσιμης αλληλείας πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος, πολυμερής προσέγγιση έχουμε αυτή τη συμφωνία του βορειοανατολικού Ατλαντικού. Κάνω όμω έκκληση υπέρ τη πολυμερού προσέγγιση και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα ενημερώσει για το τι μέτρα θα λάβει για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι μονομερεί ενέργειε ε, τη Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια. Από ό,τι κατάλαβα από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ε, υπάρχει υπεραλίευση αλλά ακούγοντα ε, αυτά που λέει ο εκπρόσωπο τη Γρυλανδία, φαίνεται πω είναι διαφορετική κατάσταση. Με την πληροφόρηση που έχω, ο Άισι είχε κάνει μία πρόβλεψη τον περασμένο Οκτώβριο για την κατάσταση των αποθεμάτων και τον περασμένο Ιούνιο μετά από έτοιμα της Νορβηγίας ακριβώς πρότειναν ε, να αυξηθεί η αλίευση κατά 100% σχεδόν. Δηλαδή, η σύσταση που είχε γίνει το προηγούμενο, το προηγούμενο φθινόπωρο αναθεωρήθηκε. Ιδιαίτερα για το σκουμπρί, λοιπόν, όπως λέγαμε. Αυτό είναι λυπηρό, γιατί αυτό είχε επίπτωση και στην κατανομή των ε, ποσοστώσεων το περασμένο χρόνο. Για παράδειγμα, ο στόλος από την Κορούνια με βάση την ποσόστοση που είχε μόνο 8 μέρες μπορούσε να ε, αλλιεύσει. Οπότε η συζήτηση αυτή μας επιτρέπει να συζητήσουμε για αυτό το λάθος στη μελέτη του ISIS. Εφόσον είναι τόσο καλύτερη η κατάσταση με τα σκουμπριά, θα ήθελα να μας πει γιατί, να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχει πρόβλημα υπεραλίευσης. Νομίζω πως αυτά τα δύο είναι αντιφατικά. Εφόσον το ISIS ε, είπε ότι έχουμε πολύ περισσότερα ελεύματα, πώς υπάρχει υπεραλίευση. Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νάβαλ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με αυτό που μόλις ε, ακούσαμε. Η σύσταση του ISIS ε, εξέπληξαν πολλούς και ιδιαίτερα τους ε, Αλής. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαπραγμάτευση που ελπίζω να επιτύχει και να τονίσω τα εξή για αυτήν. Διαπραγμάτευση με τους φίλους και εταίρους μας. Πρώτον, κοιτάξτε, Λυπάμαι που δεν ήρθε η Ισλανδία. Θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή τους. Να μας εξηγήσουν γιατί ε, υπάρχει τόση αλίευση σε διεθνή ύδατα και τόσο λίγο στα δικά τους χωρικά ύδατα. Κοιτάξτε, η υπεραλίευση είναι σημαντικό πρόβλημα. Αλλά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει θα πρέπει να δούμε πού ακριβώς αλλιεύουν τα διάφορα κράτη. Πόσο στα διεθνή, πόσο στα χωρικά τους ύδατα. Και η Ισλανδία νομίζω ότι ε, φέρεται πολύ διαφορετικά από τους άλλους θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διαπραγματεύση και να τονιστεί αυτό. Αν όλα τα παράκτια κράτη συμπεριφέρονταν με αυτόν τον τρόπο, θα είχαμε σοβαρά προβλήματα. Τώρα για την υπεραλίευση. Δεν νομίζω ότι οι ποσοστώσεις ε, του σκουμπριού είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η βιωσιμότητα του κλάδου. Αν δούμε σε τι τιμή πουλείται, πωλείται το σκουμπρί, θα καταλάβουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί η κερδοφορία του κλάδου. Γιατί όσο περισσότερα, περισσότερο σκουμπρί αλλιεύουμε, τόσο περισσότερο πέφτει η τιμή. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να κάνουμε με τους φίλους στην ε, Γρυλανδία και Ισλανδία. Κανείς δεν θα ωφεληθεί εάν ε, ψαρεύουμε περισσότερο Πουλάμε φθηνότερα και καταρρεύσει ο κλάδο. Παρακαλώ, εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, χρόνια το συζητάμε αυτό το θέμα, αλλά σας ευχαριστώ που το ξαναθέτουμε στην ημέρα στη διάταξη. Η Ισλανδία δεν παρίσταται. Χαίρομαι που παρίσταται η Γρυλανδία. Διαπιστώσαμε ήδη ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Επιτροπή είπε ότι υπάρχει 25% υπεραλίευση. Η Ιρλανδία λέει ότι αυτό δεν συμβαδίζει με τις προβλέψεις του ISIS. Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Θα πρέπει να ξαναδούμε ε, τα επιστημονικά στοιχεία. Είναι πολύ διαφορετικές αυτές οι θέσεις. Και τις ακούσαμε μέσα σε πέντε λεπτά. Οπότε, κοιτάξτε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει και ε, πώς έχουν τα πράγματα με τη Ρωσία. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τη Ρωσία, όχι μόνο με την Ισλανδία και τη Γρυλανδία. Και δεν ακούμε πολλά για τη Ρωσία. Ξέρουμε ότι τη Ρωσία έχουμε και γεωπολιτικά προβλήματα βεβαίως. Έχουμε όμως και προβλήματα στην αλλήλεια με τη Ρωσία. Να μας πει λοιπόν περισσότερα παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι θα κάνουμε για τη Ρωσία και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Πούμπεο. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγγνώμη δεν άκουσα ότι καλούσα το όνομά μου. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπο. Ναι, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Γρυλανδία που παρίσταται. Για τη στάση του νομίζω ακριβώς είναι έκφραση των λόγων του ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο για να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Γιατί η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι μέρος του προβλήματος που έχουμε για το θέμα αυτό. Λοιπόν, οι ερωτήσεις μου και έχοντας ε, ακούσει και τον εκπρόσωπο της Γρυλανδίας, η ερώτησή μου λοιπόν είναι, παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας πει γιατί όταν παρατάθηκε αυτή η συμφωνία, αυτή η τριμερή συμφωνία στην έτσι του 2014, γιατί δεν συμπεριλήφθη η Γρυλανδία που έχει ακριβώς κάθε διάθεση να συμμετάσχει. Και κάτι που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Αυτή η διαφορά μεταξύ της έκθεσης του ίσες που χρησιμοποιεί και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και ο εκπρόσωπος της Φιλανδίας. Είναι ίδια ή όχι αυτή η επιστημονική έκθεση. Δεν ξέρω πώς δεν κατάλαβα καλά, αλλά τα στοιχεία και οι προτάσεις που κάνουν ε, είναι σε εντελώ διαφορετικό σημείο. Με βάση την ίδια επιστημονική έκθεση, ο ένας λέει να μην αυξηθούν οι ποσοστώσεις και με βάση την ίδια επιστημονική μελέτη, οι άλλοι αυξάνουν την ποσόστοσή τους. Μονομερός και η Γρυλανδία και η Ισλανδία. Μα ποια έκθεση είναι και τι λέει. Πώς είναι δυνατόν να ερμηνεύεται τόσο διαφορετικά. Και Κοιτάξτε, να αναφερθώ στη δική μου κατάσταση. Η αλίευση από τους ε, Βάσκους του σκουμπριού μειώθηκε κατά 42% το 19 σε σχέση με το 18. Τι να σας πω. Δεν καταλαβαίνω. Βρίσκομαι σε κατάσταση σύγχυσης. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας πει. Σε τι στοιχεία βασίζονται. Πώς έλαβαν αυτές τις αποφάσεις ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη μία μας λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος υπεραλήψης και οι επιστημονικές εκθέσεις εφόσον υπάρχουν. Και τι προβλέπουν για του χρόνου. Θα υπάρξει ενδεχόμενη αύξηση με βάση τα στοιχεία του ISIS μετά την τελευταία αναθεώρηση. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς βλέπει το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Μοντίθ. Με εξέπληξαν. Αυτό που υπόθηκε ότι εξεπλάγει η Επιτροπή από τις αλλαγές. Είπε ότι ήταν κεραυνός ενεθρία αυτές οι αλλαγές των ποσοστώσεων. Κοιτάξτε, αυτές οι χώρες εξαρτώνται κατά πολύ από την ε, αλία για την οικονομία τους. Οπότε υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για τα επιστημονικά στοιχεία. Προσπαθούν να αλλιεύσουν το μέγιστο που επιτρέπει η επιστημονική που επιτρέπουν οι επιστημονικές εκθέσεις που λαμβάνουν. Όταν προέκυψε αυτή η τελευταία έκθεση του ISIS που επέτρεπε τέτοια τεράστια αύξηση της αλίευσης και βλέπουμε ότι και οι δύο χώρες αύξησαν ε, την αλίευσή τους λιγότερο από όσο πρότεινε η, η έκθεση του ISIS. Αυτοί ε, αύξησαν κατά 30 και 18 ενώ η ISIS η έκθεση της ISIS έλεγε ότι αυξήθηκαν τα αποθέματα κατά 100%. Ήταν λοιπόν μετριοπαθής η αύξηση αυτή. Γιατί εξεπλάγει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα τι έγινε. Το είχα ρίξει τον ύπνο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβλεψε ότι εφόσον, υπήρχε νέα, ε, εφόσον υπήρχαν νέα στοιχεία, φυσιολογικά οι δύο αυτές χώρες θα επεδίωκαν να επωφεληθούν. Πρόεδρος, ωραία. Αρκετές ερωτήσεις ετέθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλη, ε, ένα άλλο γύρο ερωτήσεων, αλλά να δώσουμε τώρα την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικές για να καταλάβετε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση, αν επιτρέπετε. Γιατί νομίζω ότι είναι βασικό στοιχείο. Ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με αυτές τις χώρες. Εξεπλάγημεν, όπως είπα, από τις αποφάσεις αυτές. Ή τουλάχιστον από το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές βασίζονταν σε εντελώς διαφορετικές παραμέτρους από ό,τι στο μέλλον. Γιατί εξεπλάγημεν. Οι δύο χώρε αυτέ συμμετείχαν στι διαβουλεύσει που έγιναν φέτο το Μάιο. Ήταν παρούσε. Και ακόμη και αν δεν ε, συμμετέχετε στη συμφωνία διανομή, όπω λέγεται, όλα τα παράκτια και ε, αλλιεύοντα κράτη καλούνται συστηματικά σε αυτέ τι διαβουλεύσει. Όλοι έχουν δυνατότητα να, εκφράσουν, να εκφράσουν την άποψή του, ιδιαίτερα για τι ε, επιστημονικέ συμβουλέ και όλες αυτές οι διαβουλεύσεις ε, ενθαρρύνονται, ε, παρακαλούνται να δώσουν ε, τις απόψεις τους για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τα θέματα του σκουμπρίου στο μέλλον. Έχουμε μια κατάσταση όπου όντως δεν είναι τέλειος ο κόσμος. Δεν έχουμε συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία όλων των παρακτήων και αλλιευών κρατών, αλλά όλοι είναι γύρω από το τραπέζι για να συζητήσουν για τη διαχείριση των αλλιευμάτων και για τι θα γίνει για αυτά τα θέματα στο μέλλον. Γιατί εξεπλάγημε λοιπόν. Γιατί σε κανένα σημείο ή οι παρόντες σε αυτές διαβουλεύσεις οι εκπρόσωποι, οι επίσημοι εκπρόσωποι των χωρών τους σε καμία χρονική στιγμή δεν έδωσαν οποιαδήποτε ένδειξη ότι δεν επρόκειτο να σεβαστούν αυτά που θα αποφασίσουν τα άλλα παράκτια κράτη και ότι επρόκειτο να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους με βάση εντελώς διαφορετικές παραμέτρους. Επαναλαμβάνω ότι εξεπλάγημεν και όχι απλώς εξεπλάγημεν, ε, δυσταστηθήκαμε ιδιαίτερα. Γιατί όχι μόνο αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση όπου τρεις εβδομάδες μετά από τις διαβουλεύσεις ενημερωθήκαμε από άλλο κανάλι για αυτές τις αλλαγές, αλλά οι παρόντες στη διαβούλευση δεν ε, ε, ε υπενήχθησαν καν ότι πρόκειτο να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Αυτό είναι, πώς να το πω, ε, είναι απίστευτο. Γιατί έχουμε σε θελούσια βάση μια διαδικασία διαβούλευσης που έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμεθα τα αλλιεύματα. Με βάση τις συμβουλές του ΆΙΣΕΣ, αναμένουμε αυτούς που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών να διατυπώσουν σαφώς τις προθέσεις τους. Και αν δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις που λαμβάνονται, αναμένουμε να εκφράσουν σαφώς την άποψή τους. Γίνανε διαβουλεύσει. Και μετά, επειδή αποφασίσαμε να υπάρξει σταθερότητα στα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα για να φτάσουμε κοντά στα μέγιστα βιώσιμα αλλιεύματα για το 2019 ήδη και όχι το 2020 μετά λοιπόν αυτές τις δύσκολες αποφάσεις στις διαβουλεύσεις ξαφνικά αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου τρία κράτη λαμβάνουν μονομερείς αποφάσεις να αυξήσουν τα λεύματά τους, να θέσουν κινδύνο αυτή την προσπάθεια, αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω ότι και εξεπλάγημεν, αλλά και απογοητευθήκαμε σφόδρα για αυτές τις ε, ενέργειες. Τώρα για τις συμβουλές του ΆΙΣΕΣ. Επανειλημμένα υπόθηκε. Πρώτα απ' όλα Κοιτάξτε, είναι δύσκολο είδος για τους επιστήμονες για να κάνουν σωστές εκτιμήσεις. Ήταν δύσκολο να υπάρξουν επαρκώς αξιόπιστα μοντέλα για να κάνουμε προβλέψεις. Αυτή τη φορά το ISIS έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να ε, βελτιώσει κατά πολύ την προσωμείωση που κάνει, ιδιαίτερα λόγω καλύτερης επεξεργασίας των στοιχείων ούτω ώστε εμεί που διαχειριζόμεθα την κατάσταση να έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε ευχερέστερα για το μέλλον. Και να πάω λίγο πίσω χρονικά. Το 2018 είχαμε τις συμβουλές του ISIS για το 19 που έδιναν μια ιδιαίτερα δεινή εικόνα μείον 61% μείωση. Πρότειναν οι επιστήμονες και ε, μείον 43% με βάση μια άλλη παράμετρο. Αλλά το ISIS κατόπιν παραδέχτηκε ότι το μοντέλο τους αυτό έπρεπε να αναλυθεί περισσότερο. Έτσι λοιπόν πέρυσι βασιστήκαμε στη γνώμη του ISIS, αλλά υπήρχε προοπτική, όπως είπα, να φτάσουμε στα μέγιστα βιώσιμα αλλιεύματα το 2020. Και αυτό το λένε τα πρακτικά, το οποίο υπογράψαμε όλοι. Τώρα όμως, φέτος, είχαμε νέες συμβουλές από το ISIS, που παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για το αλύβμα αυτό, για το απόθεμα αυτό. Και είχαμε λοιπόν μία δυσχέρεια. Θα αλλάζαμε πλήρως τα επιτρεπόματα αλλιεύματα για φέτος ή θα περιμέναμε μερικούς μήνες όταν θα συναντηθούμε για τις διαβουλεύσεις για το 20 πριν πάρουμε την απόφαση να αλλάξουμε τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση, όπως σας είπα, αλλά αποφασίσαμε ότι θέλουμε σταθερότητα. Και λαμβάνοντα αυτή την απόφαση, επίσης αποφασίσαμε να μειώσουμε ουσιοδό τα αλλιεύματα σκουμπριού. Και το είπα και νωρίτερα, ότι θέλουμε να αλλάξουμε κατά λίγους, λίγες ποσοστιαίες μονάδες. Τα, παρελθόντα έτη είχαμε φτάσει σε υπεραλίευση μέχρι και 25%. Μέσω της απόφασης να μην αλλάξουμε τα ΤΑΚ και αν τα τρία αυτά κράτη, Ισλανδία, Γρυλανδία και Ρωσία, είχαν αποφασίσει να μην αλλάξουν την ποσόστοσή τους, τότε το απόθεμα θα ήταν πολύ κοντά στο βιώσιμο ήδη από το 2019. Στο μέγιστο βιώσιμο αλλήλωμα. Αυτός ο στόχος υπονομεύεται από τις μονομερείς αυξήσεις ποσοστώσεων αυτών των τριών κρατών. Εδώ είμαστε τώρα. Και όσον αφορά τη Ρωσία, γιατί τέθηκε. Δεν ε, μεταχειριζόμεθα διαφορετικά τη Ρωσία. Η Ρωσία απέχει στο παρελθόν, απήχε για τα τελευταία δύο χρόνια των διαβουλεύσεων. Και πρόσφατα έχουμε δυσκολίε για να βρούμε ε, τρόπο επικοινωνία με τη Ρωσία. Θα του δούμε τι επόμενε εβδομάδε. Θα υπάρξουν περαιτέρω διμερείς επαφέ μεταξύ των άλλων παρακτήων κρατών και τη Ρωσία. και υπάρχουν κάποιε ενδείξει πολύ πρόσφατα ότι δεσμεύονται να συμμετέχουν στο μέλλον σε όλε τι διαβουλεύσεις και ιδιαίτερα αυτές που θα γίνουν τον προσεχή Οκτώβριο για το Σκουμπρί, για τη Ρέγκα και ένα άλλο είδος για το 2020. Είπαμε επίσης ότι θα στείλουμε μία παρόμοια ανακοίνωση στη Ρωσία με αυτή που στείλαμε στην Ισλανδία και την Ιρλανδία αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο να συνεργαστούμε μαζί τους γιατί δεν έχουμε καν ε, εύκολα δυνατότητα να έχουμε διάβολο επικοινωνία με τη Ρωσία. Και τέλος, προοπτικές μέλλοντος. Τέθηκε το ερώτημα. Κοιτάξτε, είναι λίγο νωρίς. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκα σε μια τεχνική ομάδα εργασίας, συναντήθηκαν σε μια τεχνική ομάδα εργασίας οι επιστήμονες για να δουν και τα στοιχεία και το μοντέλο που θα διαμορφώσουν τις συμβουλές που θα λάβουμε σε μερικές εβδομάδες για το 2020, τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι πολύ διαφορετικές συμβουλέ τους από αυτέ που λάβαμε για φέτος, αλλά δεν θέλω να προκαταλάβω τις συζητήσεις. Ας αφήσουμε τους επιστήμονες να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους που να είναι επαρκώς αξιόπιστες γιατί εμείς πρέπει να λάβουμε με βάση τα στοιχεία αυτά τις αποφάσεις διαχείρισης. Γι' αυτό ας τους αφήσουμε χρόνο να κάνουν ε, μια εκλέπτυνση των ε, συμβουλών τους. Εγώ δεν έχω αυτά τα στοιχεία τώρα για το προς τα που πάει η κατάσταση, δεν ξέρω αν τα έχετε εσείς. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όπως σας είπα, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου αναμένουμε αυτές τις συμβουλές και κατόπιν θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία που θα μας επιτρέψει να λάβουμε τις αποφάσεις μας για τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα το 2020. Ας περιμένουμε λοιπόν τη γνώμη του ΆΙΣΕΣ πριν ε, αποφασίσουμε το μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Δονατέλα, Θα έπρεπε να σας πω ότι έχω έρθει σε επαφή με εκπροσώπους ε, Βρετανών και Ιρλανδών αλλιών τις περασμένες εβδομάδες, 75% δηλαδή ε, του αλλιεύματος ε, σκουμπριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άσκησαν ε, κριτικές αρνητικές στην Κομισιόν γιατί είπαν ότι επέτρεψαν στην Ισλανδία και την Ισλανδία αλλά κυρίω την Ισλανδία να κάνει ό,τι θέλει. Με σχεδόν, από σχεδόν μηδενικό αλίευμα τώρα φτάνει στους 140.000 τόνου, από τους οποίους 60% προέρχεται εκτό των χωρικών του υδάτους. Είπαν ότι η Κομισιόν έδειξε δυναμία και ότι ε, θυσίασε τα δικά του συμφέροντα ώστε να μπορέσει να φτιάξει μια επόμενη συμφωνία για τους 12 μήνες που έρχονται. Πολλές επικρίσεις λοιπόν. Έχω έρθει επίσης σε επαφή με εκπρόσωπους της Ισλανδίας. Μάλιστα αυτό έγινε χτες. Που ε, βεβαίω παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα και λένε ότι ε, τονίζουν ότι θέλουν μια επίσημη συμφωνία με τις νήσους Φαρόε, την Νορβηγία και την Ένωση, ότι θα πρέπει να είναι πιο μακροχρόνια συμφωνία, ότι θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και του σεβασμού για τις συμβουλές του ΆΙΣΕΣ και βεβαίως ε, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεπής ε, και οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι συνεπής στο συμβουλές του ISIS και θέλουν να μπορούν να έχουν το μερίδιο σκουμπριού που τους αναλογεί. Είναι έτοιμοι να αρχίσουν να συζητούν όχι από το νούμερο που τώρα συζητούν, το 21,5 1% αλλά το, 12% ε, που ισχύει όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει το 2014. Τελείω διαφορετική θέση λοιπόν. Και είμαι βέβαιο βέβαιος ότι η Επιτροπή θα πρέπει προκαταρχά για να κλείσει μια συμφωνία να προστατεύσει τα συμφέροντα των δικών μα αλλιέων αλλά και να υπάρχει να εξασφαλίσει την ύπαρξη βιώσιμου αλλιεύματο κουμπριού για το μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ίσως ε, το ισχυρότερο μέσο που έχετε, δηλαδή κυρώσεις μάλλον, για να μπορέσετε να φέρετε τον κόσμο στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Ίσως όμως υπάρχει και κάποια προθυμία για διαπραγμάτευση και αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε βέβαια και ο Ισλανδός εκπρόσωπος ε, μίλησε για εμπιστοσύνη και να πούμε λοιπόν και εμείς ότι ε, εφόσον αυτό θέλατε και εμείς αυτό επιθυμούμε ε, και μήπως θα πρέπει να διερευνηθούν και άλλα θέματα, ας πούμε το θέμα του Σιρέγκας και άλλων ειδών και μήπως δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη, βρύτερη συμφωνία με αυτά τα είδη και με το μερίδιο σκουμπριού. Θέλετε να το σχολιάσετε? Σας ευχαριστώ πολύ. Και όντως είναι περίπλοκη η κατάσταση α, όπως την περιγράψατε. Ε, σίγουρα στο πεδίο του Σκουμπριού εστιάζουμε σε αυτό το θέμα γιατί είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν είναι το μόνο και, ότι ενός, και βεβαίως ε, εν, συζητάμε ε, το Σκουμπρί, συζητάμε και την Ρέγκα και τον Ταούκι. Ε, και μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όντως σε μια συμφωνία, αλλά ούτε αυτό έχει φανεί εύκολο. Είναι ζήτημα λοιπόν για το σκουμπρί, αλλά όχι μόνο. Και ενώ εστιάζουμε στο συγκεκριμένο είδος, ε, ε, είναι προς το συμφέρον μας να δείξουμε πως έχουμε ευρεία και καλή σχέση με τους βόρειους μας εταίρους αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν ε, ε, ταγκό, δύο για να συνάψουν μία ε, συμφωνία και αν οι εταίροι δεν εμφανίζονται σε συνεδριάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά όσον αφορά τη συνέχιση αυτής της σχέσης. Επόμενη η συνεδρίαση προβλέπεται για τον Οκτώβριο. Όλοι έχουν προσκληθεί και ελπίζω πως όλοι θα εμφανιστούν γιατί είναι πολύ σημαντική η συμφωνία αυτή για αυτά τα αλληλευτικά αποθέματα. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να μας πείτε τι έγινε σε αυτή τη συνεδρίαση μετά. Θέλετε να πείτε τώρα εσείς κάτι, κύριε Κλάς, για την επόμενη, ε, για τη λήξη μάλλον αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε καταρχάς. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε να δώσουμε τη γνώμη μας. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε με τη συνεργασία και πραγματική πολυμερή συμφωνία όπου δηλαδή όλα τα παράκτια κράτη θα είναι μέρη της ε, ε συμφωνίας για το Κουμπρίπρους Βλέπουμε στις επόμενες διαπραγματεύσεις για μια μελλοντική συμφωνία όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και όπου θα υπάρχουν ωφέλη για, ε, για όλους. Σε ένα λοιπόν ε, πνεύμα συνεργασίας, ναι, ας το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Ντονατέλα και του συναδέλφου, σα Είμαι βέβαιος πώ θα επανέλθουμε στο θέμα και θα, σας, θα τα ξαναπούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο επόμενο σημείο και καλωσορίζουμε τον Υπουργό της Φιλανδίας. Very well, thank you. Could you take your seats, please? Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Καθίστε παρακαλώ. Λέπε, λέπε, λέπε, λέπε, It's yes. yes. Yes, of course. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Ε, ε, ξεκινάμε. I'd like Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάρη Λέπε που είναι υπουργός ε, για τα δάση των δασών στην Φιλανδία καλύπτει και την Αλία. βέβαια ήδη έχει μισοτελειώσει η Προεδρία. Εν μέρει έχουμε καθυστερήσει γιατί ο υπουργό μου έδειχνε μια εικόνα του μεγαλύτερου ψαριού που έχει ποτέ ψαρέψει. 10 κιλά ψάρι έπιασε, σχεδόν το μέγεθο της κόρη του. Του έλεγα ότι το Photoshop ε, λειτουργεί πολύ καλά τη σήμερα ημέρα και ότι μπορείς να κάνεις διάφορα ωραία με τα μεγέθη των ψαριών. I can give you an introduction, but I, th I, think, I think the floor is yours. Αρκετή εισαγωγή έκανα. Ε, μπορείτε να πάρετε εσείς το λόγο τώρα. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Meillä on... Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, μέλη τη Επιτροπή, είναι τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τη Φιλανδική Προεδρία. Πρώτα απ' όλα εξ αρχής θα ήθελα να πω και να τονίσω πόσο πολύ σημαντικό είναι για μένα προσωπικά να διεξάγω διάλογο ο οποίος προάγει την ε, αγαστή συνεργασία μεταξύ των ε, θεσμών ώστε να προοδεύσουν τα θέματα που αφορούν την αλληλεία. Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξέλεξαν ως εκπροσώπους τους πρόσφατα και θέλω να σας συγχαρώ όλους εξ αρχής. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εργασία σας. Εκτιμώ πολύ τη δουλειά που κάνετε εδώ στην Επιτροπή σας, διότι παίζετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορείτε να υπερασπίσετε τα συμφέροντα των πολιτών και το... της αλληλείας και να υπερασπιστείτε τις κοινέ ευρωπαϊκές αρχές. Η σημερινή επαφή είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της ε, προσήλωσής μας ε, και του ανοιχτού πνεύματος που θέλουμε να επιδείξουμε στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας. Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι κύριοι ευρωβουλευτές, θέλω να πω καταρχάς δύο λόγια για τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Στη συνέχεια θα μπω πιο εις βάθος σε θέματα που εμπίπτουν στην εντολή της Επιτροπής σας. Σε σχέση με την Φιλανδική Προεδρία και το πρόγραμμά μας, Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να προωθήσουμε τον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών και τον σεβασμό ε, των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον θα θέλαμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια, την σταθερότητα και να καταστήσουμε πιο συνεκτική την Ευρώπη από κοινωνική άποψη. Οι κατευθυντήριε γραμμέ είναι λοιπόν το ανοιχτό πνεύμα, η εμπιστοσύνη, η χρηστή διαχείριση και η βιωσιμότητα. Στον ε, επιτάπητος υπήρχαν πολλά κρίσιμα θέματα όσον αφορά το μέλλον της Ένωσης και την εξέβρεση λύσεων. Ε, θα πρέπει καταρχάς να βρούμε σωστή ισορροπία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι καλύπτει τα παραδοσιακά μας μέσα αλλά και τις νέες προκλήσεις. Το επόμενο PDP θα, θα ε, επηρεάσει σίγουρα και την κοινή αλληλευτική πολιτική. Όσον αφορά την αλληλεία, η Φιλανδική Προεδρία θα έχει πολλή δουλειά μπροστά της Καταρχά, θα ήθελα να τονίσω ότι η αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς καθώς και η προσήλωση στους στόχους της, κοινή αλευτικής πολιτικής καθώς και η χρήση των πιο πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων μας βοηθούν στο να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους και για τους αλληλείς και για τα αλλιεύματα και για τους καταναλωτές. Όσον αφορά τις τα μεγαλύτερα επιτρεπόμενα αλλιεύματα και τις ποσοστώσεις, θα πρέπει να σας πω ότι τα μέτρα αυτά έχουν συμβάλει στη θετική εξέλιξη για πολλά από τα αποθέματα που έχουν σημαντικά αυξηθεί και διαχείρισή τους γίνεται επί τη βάση της μέγιστης ε, ε, βιώσιμης ε, απόδοσης MSY. Παρά όμως τις προσπάθειες, τα αποθέματα βακαλάου έχουν μειωθεί σημαντικά ε, και θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα εκεί. Τώρα, τα τάκ και οι ποσοστώσεις για τη Βαλτική θάλασσα, για τη Μαύρη θάλασσα, τη Βόρεια θάλασσα και το Βόρειο Ατλαντικό θα οριστούν επίση στη διάρκεια της Προεδρίας μας και για πρώτη φορά αναμένουμε η Επιτροπή να μας υποβάλει πρόταση για την ε, μέγιστη επιτρεπόμενη αλληλευτική προσπάθεια και στη Μεσόγειο. Εμείς ε, ε, πιστεύουμε στην βιώσιμη διαχείριση των ελευθερικών αποθεμάτων και ελπίζουμε ότι μέχρι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε επιτύχει ένα από τους κεντρικούς στόχους της ελευτικής πολιτικής, δηλαδή τη μέγιστη ε, βιώσιμη απόδοση. Δουλεύουμε πολύ στενά με όλα τα ε, εμπλεκόμενα κράτη-μέλη και την Κομισιόν, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση θα ε, εξασφαλιστεί για το 2020 και θα συμφωνηθεί μεταξύ όλων των πλευρών. Όπως γίνεται κάθε χρόνο θα σεβαστούμε τις αρχές και του στόχους της κοινή αλευτικής πολιτικής, δηλαδή και την λήψη αποφάσεων επί τη βάση ε, των πιο έγκυρων επιστημονικών συμβουλών και δεδομένων. Έχουμε σχέδια για διάφορα επίπεδα, για διάφορα μάλλον διάφορες θαλάσσιες περιοχές, χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε βιώσιμα τα αλληλευτικά αποθέματα. Αναμένουμε ότι φέτος η κατανομή των ποσοστώσεων και των ΤΑΚ ε, θα είναι μια δύσκολη διαδικασία σε συνδυασμό με την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, γιατί υπάρχουν διάφορες αβεβαιότητες. Υπάρχει ο αντίκτυπος ε, που είναι αδύνατο να εκτιμήσουμε σε αυτή τη φάση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτές οι αβεβαιότητες και φυσικά θα τις λάβουμε υπόψη όπως πρέπει. να πω και δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας και ε, Θαλασσών. Πρόκειται για ένα θέμα που συνδέεται στενά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που είναι ένα σημαντικό μέσο για, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιδευθούν οι στόχοι της κοινή αλευτικής πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα όσο περισσότερο γίνεται στη διάρκεια της Προεδρίας και ελπίζουμε πώς θα ε, μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια μερική κοινή θέση στην ε, ε, συνεδρίασή μας του Οκτωβρίου για τη Γεωργία και την Αλία. Ε, και ε, πιστεύουμε πως έτσι θα μπορέσουμε ε, να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και στους τριμερείς διαλόγους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο κάνει μια λεπτομερή ανάλυση της πρότασης της Κομισιόν που σχετίζεται με τον έλεγχο το, της αλληλείας ε, η ιδέα είναι να ενημερωθεί και να ανανεωθεί η νομοθεσία περί ε, ελέγχων. Ε, η ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτό είναι να απλοποιηθούν οι κανόνες ώστε να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το φόρτο τόσο του διοικητικού μηχανισμού όσο και των αλλιέων και της αλλιευτικής βιομηχανίας. Και εκεί προσπαθούμε να το προχωρήσουμε όσο γίνεται μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Ως προς αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η Φιλανδία εξετάζει πολύ σοβαρά το θέμα της υπεύθυνης αλληλείας. Ε, ε, αγωνιζόμαστε πολύ σκληρά κατά της παράνομης αλληλείας γιατί είναι βλαβερή για τη βιωσιμότητα των αλλιευμάτων. Επίσης είναι σημαντικός ο αγώνας αυτός για την εγγύηση της ίσης μεταχείρισης ε, των αλλιέων αλλά και όσον αφορά την δικαιοσύνη γιατί οι αλληλείς που ακολουθούν τους κανόνες δεν θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν από το γεγονός ότι δεν παίζουν όλοι με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού. Ως προς αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και παίζει ε, σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, οι περιφερειακές ε, οργανώσεις διαχείρισης των αλλιευμάτων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί βοηθούν στην ε, συνεννόηση και στην ε, προώθηση, της βιώσιμη προώθηση μάλλον, των αλευμάτων. Οι περιφερειακές οργανώσεις αλίες καθώς και οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα το, της αλίες είναι θέματα τα οποία απασχολούν την Φιλανδική Προεδρία και στα οποία θα επιτείνουμε τις προσπάθειές μας. Θα ήθελα λοιπόν εδώ και πάλι να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, μιλήσω σήμερα και προσβλέπω στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ακολουθήσει και στις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κατανοούμε βεβαίως όλοι ότι έχετε την ευθύνη στο Συμβούλιο να καταλήξετε σε συνένεση και να προχωρήσετε σε πολλά θέματα. Αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε στην Επιτροπή μας εσείς κατά πόσον μπορείτε με τον ενθουσιασμό σας να επηρεάσετε και τους συναδέλφους σας, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν κάποιοι από τους στόχους σας στο Συμβούλιο. Θα το δούμε. Ο κύριος Μιλανμόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ήρθατε να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Ξέρουμε ότι είναι πολύπλοκο αυτή η εποχή. Σας εύχομαι ε, για τα ποσοστώσεις και τα τάξη επιτυχία. Τώρα το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου όχι μόνο την ε, βιωσιμότητα ε, για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα, κυρίως τον τομέα της αλίας και νομίζω ότι και αυτή τη διάσταση και εσείς την έχετε συμπεριλάβει προτεραιότητας όσον αφορά επί της ουσίας. Χαίρομαι που είναι ε, ε, προτεραιότητα για σας όπως και για μας όταν τον Απρίλιο ε, αρχίσαμε να κάνουμε τις διάφορες δίσεις τα πέσια του τριμερούς διαλόγου για το ταμείο το και θέλουμε να έχουμε ένα ταμείο με τους απαραίτητους πόρους. Δεν θέλουμε να υπάρχουν ε, κυρίως περικοπές και να είναι η δικαιολογία του Brexit μια άριστη δικαιολογία για να μπορέσουν ε, τα κονδύλια που προβλέπονται για το ταμείο να μειωθούν. Θα ήθελα να υποφεληθώ τη παρουσία σας κύριε Υπουργέ για να επιμείνω πόσο σημαντικές είναι οι αλληλευτικέ συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ε, βιώσιμης αλίας θα ήθελα να πω. Κατά την ε, διάρκεια προεδρία σας, εάν είμαι καλά ενημερωμένο το Νοέμβριο εκπνέει η συμφωνία με την Μαυριτανία. Είναι πάρα πολύ σημαντική, ίσως η πιο σημαντική που έχουμε σήμερα με κάποια από τις τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να προσέξει αυτό το θέμα. Και για να μπορέσουμε να κάνουμε μία σωστή, αποτελεσματική και ήρεμη διαπραγμάτευση, ίσως θα πρέπει να ζητήσετε ε, και παράταση ενός έτους, ώστε να μην γίνουν ε, βιαστικά κάποια θέματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσετε και εσείς με την Κομισιόν το θέμα που υπάρχει από το Μάρτιο στα βόρεια ε, σύνορα της ε, Μαυριτανίας που εμποδίζουν τη διέλευση κάποιων πλοίων. 11 από αυτά προέρχονται από τη δική μου περιοχή, τη Γαλλικία. Υπάρχουν λοιπόν μπλοκάρι η είσοδό του και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται και κάτι το οποίο δημιουργεί τρομερά προβλήματα και επιδεινώνει την κατάσταση του δικού μα αλληλευτικού στόχου. Θα ήθελα να το προσέξετε ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Δεν είναι και ελάσσονο σημασία. Κάθε μέρα, τουλάχιστον στη δική μου περιοχή, στη Γαλλική, εμφανίζονται τέτοιου είδου σχόλια για το θέμα αυτό κάθε μέρα. Στι 28 Αυγούστου, επίσης, στον τύπο εμφανίστηκε το περίφημο θέμα του Καρχαρία Μαράχο, όπως το λέμε εμείς. Με προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά των επιστημονικών συστάσεων και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προηγούμενο. Στο... Η συμπερίληψή του στο παράρτημα 2 δεν εγκρίθηκε ούτε από τη γραμματεία της ΦΙΤΟΣ ούτε από τη ΦΑΟ. Πρόκειται για ένα είδος το οποίο χειρίζονται οι όροπες πολύ καλά. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει πρόβλημα ε, εξάντλησης των αποθεμάτων. Και η απόφαση αυτή εξέπληξε την, ε, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε αυτής της αποφάσεις του Μεξικού. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε γιατί εγκρίθηκε μια τέτοια απόφαση εάν ελήφθη όχι από τους ε, υπουργούς αλίας αλλά ίσως από τους υπουργούς περιβάλλοντος ή τους υπεύθυνου για την γεωργία και την αλία. Το γνωρίζουν αυτό το θέμα. Χρησιμοποιήθηκε, λοιπόν δημιουργήθηκαν τρομερά σχόλια και πρέπει να σας πω ότι ίσως αυτό το θέμα δημιουργεί πραγματικά προηγούμενο. Τελειώνω, Πρόεδρε. Κατά συνέπεια, αυτό το προηγούμενο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιμών έθεσε πολλά ερωτήματα. Μερικά από αυτά είναι εντελώ νέα. Ίσως είναι νέα αυτά που ακούτε. Μπορείτε να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. As I Όπως σας είπα, είστε υπουργό Γεωργίας και Αλίας. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε σχέση με τις πρώτες ερωτήσεις για τα θέματα βιωσιμότητας. Η βιωσιμότητα είναι από πάσα άποψη οικονομική, οικολογική, νομική. Αυτό είναι ένα σύνολο της βιωσιμότητας και για μας είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θέλει να τονίσει η Φιλανδία ότι θα ευρεθεί λύση στα πλαίσια του MFF, δηλαδή του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Είπα πολλές φορές ότι υπάρχουν στόχοι για τις εταιρείες, για τα άτομα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχουμε ίσως και λυσμό. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες ανισοπρίες. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέγω από καιρό. Και βεβαίω αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων παίρνουν τελευταία απόφαση. Το είπα αυτό και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει όλους τους τομείς της πολιτικής. Πιστεύω λοιπόν θα μπορέσουμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία τρίτες χώρες τώρα. Συμφωνίες με τρίτες χώρες. Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι σημαντικό στα πλαίσια της εντολής του να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις για το νέο πρωτόκολλο με τη Μαυριτανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγκρίθηκε ως απόφαση πολύ πρόσφατα. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης τις ε, διαπραγματεύσεις της Επιτροπής και η προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί η συμφωνία αυτή, διότι όντως αυτό είναι προς συμφέρος του αλλιευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Τώρα, Υπάρχουν και προτεραιότητες για τους ε, υπουργούς περιβάλλοντος, για τις αρμοδιότητές τους. Δεν μπορώ να απαντήσω. Θα πρέπει να θέσετε το ερώτημα στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Μισό λεπτό. Δεν σας πω, για το θέμα της σύμβασης θήτες, αυτό το είδος καρχαρία είναι κάτι το οποίο πωλείται. Χιλιάδες τόνοι το χρόνο αλλιεύονται. Οπότε δεν είναι θέμα ε, περιβαλλοντικό μόνο. Είναι θέμα εφαρμογής των ε, συμφωνιών για την αλληλεία. Βεβαίω είναι και περιβαλλοντικό θέμα, αλλά πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς. Τονίζω, πωλείται και με βάση τα επιστημονικά στοιχεία δεν κινδυνεύει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε της ε, Φινλανδικής Προεδρίας. Να αναφερθώ και εγώ στη σημασία που θα έχει κατά τη θητεία σας η έγκριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο ουσιώδη θέματα που μας απασχολούν Πρέπει να υπάρξει η σωστή ισορροπία στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Όπως ξέρετε όμω είναι μικρό ταμείο, πολύ μικρό. Δεν ξέρουμε πως είναι το μικρότερο από πλευράς ε, πρικοδότησης από όλα τα ταμεία της Ένωσης. Οπότε να προταθεί οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή, τι έννοια έχει. Οποιαδήποτε περικοπή σημαίνει μεγάλο τμήμα. Επίσης ε, θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη της ε, γαλάζιας οικονομίας των ωκεανών. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξουν περικοπές. Και συμφωνώ ως ομάδα και με την ομάδα του κυρίου Μιγιάν Μον ότι θέλουμε και θα εργαστούμε ούτω ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή του Ταμείου αυτού και το Κοινοβούλιο θα αγωνιστεί για το θέμα αυτό και στη Γεωργία. Αλλά αυτό θα το δούμε σήμερα το απόγευμα που θα συζητήσουμε και για θέματα γεωργίας. Είναι λοιπόν ε, κυρίαρχη προτεραιότητά μας. Το, βέβαια πάντα, το βέβαιο θέμα, όπως κάθε χρόνο βέβαια, είναι το θέμα των ποσοστώσεων και των μεγίστων επιτρεπόμενων αλλιευμάτων. Και θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα εάν ε, προβλέπετε κάποια λύση για τα θέματα του βακαλάου της Βαλτικής. Ξέρω ότι είναι δυσχερές. Έχετε όμως κάτι να μας πείτε. Επίσης, τι γνώμη έχετε ως Φιλανδία, ως Προεδρία για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να εστιάσουμε περισσότερο και πιο ενιαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ψυχαγωγική αλία. Τι δυνατότητες ε, προσφέρει στα κράτη. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει να έχουμε μια πιο ομοιόμορφη αντίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτή την ψυχαγωγική αλλήλεια. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Ξέρω ότι είναι και αυτό δυσχερές θέμα. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν πολλές, ε, πολλοί δισταγμοί. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε ενιαία προσέγγιση θα πρέπει να το συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι η συγγήτρια του κανονισμού για τον έλεγχο της αλίας. Θέλουμε να υπάρξει απλούστευση. για να επιτύχουμε τους στόχους της κοινή ελευτική πολιτικής. Θα προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Χρειάζεται να αλλάξουμε εισηγητή μετά τις ε, ευρωεκλογέ, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο γίνεται και στο Κοινοβούλιο και ελπίζω και στο Συμβούλιο. Κατά λίγο, Πρόεδρε. Εμπορικές συμφωνίε. Επίση πολύ σημαντικέ. Ιδιαίτερα με τη Μαυριτανία Ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με το Μαρόκο, αλλά έχουμε και το θέμα με τη Γουινέα Μπισάου. Αυτέ οι συμφωνίε είναι πολύ σημαντικέ για τον ευρωπαϊκό στόλο. Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια, ούτω ώστε οι ψαράδε μα να εργάζονται υπό καλύτερε συνθήκε. Σα καλώ λοιπόν, όπω υπόθηκε και για τη Μαυριτανία, να προχωρήσουμε και ε, σε συμφωνία με τη Γουνέα Μπισάου, για την οποία συμφωνία ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήξερα ότι θα μου θέσετε δύσκολα θέματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τη γενικότερη εικόνα για τον Μπακαλιάρο. Από πλευράς βιωσιμότητας και με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που πρέπει να είναι η βάση της ε, σκέψης μας. Λάβαμε πρώτες προτάσεις λοιπόν με βάση αυτά που προανέφερα. Τις εξετάζουμε. Έχουν διεξαχθεί συνομιλίες με τα κράτη-μέλη, με διάφορους οργανισμούς και φορείς και μεταγενέστερα θα κάνουμε προτάσεις για τα θέματα αυτά, για, τον, ε, για τις ποσοστώσεις, για το βακαλάο της Βαλτικής. Λοιπόν, ξέρουμε ότι το απόθεμα αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα. Τώρα, ψυχαγωγική αλληλεία. Κοιτάξτε, η κατάσταση από τη μία περιοχή στην άλλη των θαλασσών μας είναι πολύ διαφορετική. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολλές αναλύσεις για να δούμε εάν και κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση σε όλες τις χώρες, αλλά είναι τόσο διαφορετικές οι διάφορες περιοχές που είναι δύσκολο να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία έχουμε τις ε, λίμνες μας οι οποίε παγώνουν το χειμώνα, ενώ σε άλλε χώρε δεν παγώνουν. Οπότε η βιωσιμότητα ε, αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Είναι δυσχερέ πολύ αυτό το θέμα. Και τα κράτη-μέλη έχουν κάποιε ευθύνε για τα θέματα αυτά. Με συγχωρείτε κάτι πολύ ε, ταχές. Αν μπορούμε να έχουμε στοιχεία, ουσιώδη στοιχεία, πραγματικά στοιχεία, αξιόπιστα για την ψαγωγική αλλήλεια. Γιατί βεβαίω υπάρχουν πολλέ ιδιαιτερότητε. Ε, έχετε δίκιο. Δεν είναι παντού οι ίδιε οι καταστάσει. Βέβαια, η κατάσταση στη Φιλανδία δεν είναι όπω στην Ισπανία. Αν μπορούμε όμω να προχωρήσουμε τουλάχιστον στη συλλογή αξιοπίστων στοιχείων για την ψαγωγική αλληλεία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ξέρετε ότι προσπαθώ να δίνω δυνατότητα να λάβουμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις, όχι γενικόλογες. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι με τις ερωτήσεις σας, ούτως ώστε να προλάβουμε να έχουμε και συγκεκριμένες απαντήσεις επί των επιμέρους θεμάτων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Μπιλμπάο. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ε, Φινλανδικής Προεδρίας. Τώρα για αυτό το ταμείο θα είναι από τα πιο σημαντικά θέματα κατά αυτή τη θητεία. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση τώρα για την αλία μας. Πολύ σημαντική μείωση των αλευμάτων σε πολλές περιοχές. Και γι' αυτό το Ταμείο αυτό θα πρέπει να βοηθήσει να βελτιωθεί και η αλία και να υπάρξει και αναγκαία διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας στις παράκτες περιοχές και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με τη βοήθεια της Ένωσης. Δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι ένα θέμα που εκκρεμεί. Τι γνώμη έχετε και αν σκέφτεστε να εξετάσετε το θέμα της απέτησης ανιχνευσιμότητας των αλληλευτικών προϊόντων. Το Κοινοβούλιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί με βάση τα προβλήματα που προκύπτουν προχωράμε για να έχουμε την ε, ηχνηλασιμότητα των διαφόρων προϊόντων για διάφορα προϊόντα, όπως για παράδειγμα το κρέας και το γάλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τα προϊόντα της αλίας. Πρώτα απ' όλα πρέπει αυτό να σημαίνει ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα του καταναλωτή να ξέρει τι αγοράζει και πόσα πληρώνει. Και θα επιτρέψει σε πολλούς τομείς της αλίας που δεν έχουν πολύ μεγάλες ποσοστώσεις να προωθήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους που είναι πολύ ε, βραχίας αλίευσης και είναι σε ε, ε, μικρό, είναι αλία μικρής κλίμακας και βιώσιμη. Για το Ηνωμένο Βασίλειο είπατε ότι θα καθορίσετε τη θέση σας. Αλλά, συγγνώμη, συγγνώμη για, την, για τη Μεσόγειο. Υπάρχει ε, ένα σχέδιο για τα αλλιεύματα Δεν κατάλαβα, θα αναφερθήκατε στα ΤΑΚ τα μέγιστα επιτρεπόμενα λιεύματα και ένα μόνιμο θέμα που θέτει το Κοινοβούλιο είναι να γίνεται σεβαστή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και η Επιτροπή Αλίας θα πρέπει να μπορεί να κάνει προτάσεις, συγγνώμη, να εκφραστεί για τα θέματα των ΤΑΚ και των αποθεμάτων έχοντα πλήρη πρόσβαση στα επιστημονικά στοιχεία, βεβαίω ξέρουμε ότι το Συμβούλιο τελικά θα πάρει την απόφαση. Θα προωθήσετε αυτή την ε, διαφάνεια που είναι και θέμα σεβασμού των αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή Αλληλεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. για την εχνηλασιμότητα. Να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Εδώ και 20 πάνω κάτω χρόνια είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η εχνηλασιμότητα είναι ένα θέμα που προωθώ μόνιμα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Για διάφορους λόγους. Και ένας λόγος είναι ακριβώς ότι οι καναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι καταναλώνουν. Και επίσης έχουν δικαίωμα να επιλέγουν τι θα καταναλώσουν. Για να κάνουν αυτή την επιλογή πρέπει να γνωρίζουν από πού προέρχεται το κάθε τρόφιμο. Αλλά το θέμα αυτό θα βοηθήσει και τους, κατανα... και τους παραγωγούς συγκεκριμένα, τους αλείς. Και αυτοί πρέπει να ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Ο πρόεδρος και άλλοι ανέφεραν ότι η πληροφορία είναι πολύ σημαντική για να κάνει τις σωστές επιλογές. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στον καταναλωτή και όσον αφορά την ίχνη λασιμότητα. Των τροφίμων πάντα και φυσικά και τα αλλιευτικά προϊόντα είναι τρόφιμα. Τώρα, τώρα τον κανονισμό για τον έλεγχο της αλίας. Ο κανονισμός αυτός θα είναι δεσμευτικός για την αλληλεία και τα αλληλευτικά προϊόντα. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να σέβονται τους κανόνες. Και έχουμε και δυνατότητες και μέσα για να επιβάλλουμε το σεβασμό των κανόνων. Και όταν θα παραστώ στην ε, ακρόαση της Επιτροπής Γεωργίας, το θέμα αυτό είμαι σίγουρος ότι θα τεθεί. Τώρα όσον αφορά τα ΤΑΚ, τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Η προσέγγιση μας, όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, είναι ότι θέλουμε καλές σχέσεις μεταξύ των θεσμών. Και κάθε θεσμός πρέπει να σέβεται και να περιορίζεται στις αρμοδιότητες ε, που έχει με βάση τις συνθήκες. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο αφετηρίας. Τώρα, για τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα, επιτρεπόμενα αλλιεύματα, θα μας απασχολήσει πολύ σοβαρά στα πλαίσια της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των θεσμών, γιατί είναι για μας πολύ σημαντικό ούτω ώστε οι αποφάσει μα να είναι πιο συνενετικέ και προ το συμφέρον γενικά τη Ευρώπη, να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι η Ευρώπη παραμένει ανταγωνιστική και ότι θα βελτιωθεί η ευημερία των συμπολιτών μα, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο την τόσο δυσχερή που διανύουμε. Η Φιλανδική Προεδρία θα ασχοληθεί και θα προωθήσει ιδιαίτερα τα θέματα αυτά. Θέλουμε σταθερή πολιτική, σταθερότητα για την κοινωνία μας. και επίσης ένα σταθερό πλαίσιο για την οικονομική μας δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνει και τους γεωργούς και την αλία γιατί υπήρξαν πολλές διαταράξεις ε, την τελευταία περίοδο. Θέλουμε λοιπόν να ενισχυθεί η σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Οσάλιβαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Σε εύχομαι κάθε επιτυχία κατά την θητεία σας. Εμείς ως πράσινοι χαιρετίζουμε τη σημασία που αποδίδεται στη βιοπικιλότητα και την βιωσιμότητα. Αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή. Και εδώ πολύ θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πρωτοπόρα όσον αφορά τη διαχείριση των ελευτικών πόρων σε σχέση με τις προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, κατά τη θητεία σας, να τοποθετήσετε την αλληλεία στο ίδιο επίπεδο με τη δασοκομεία και τη γεωργία. Τα δύο μεγάλα θέματα είναι τα ΤΑΚ για το 2020 και πώς θα δεμηθούν οι πόροι του Ταμείου Αλίας. Το 2013 εγκρίναμε την κοινή αλληλευτική πολιτική. Ήδη λοιπόν από το 2013 ελπίζω λοιπόν να τηρήσετε τις προθεσμίες και να επιτύχετε τους στόχους της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Μας ενδιαφέρει επίσης ε, η κατανομή των επιδοτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, εγκρίνει την εντολή της για την συζήτηση στα πλαίσια του ΠΟΕ για τις ε, επιδοτήσεις και έχει δεσμευθεί να καταργήσει επιδοτήσεις που δημιουργούν υπεραλίευση και που προωθούν την παράνομη, παράτυπη και ανεξέλεκτη αλληλεία. Θα πρέπει να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν τις επιδοτήσεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε εμά την Ένωση σε υπεραλίευση και υπερβολικό δυναμικό αλίευσης. Και πώς θα ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εγκρίνει τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης ιδιαίτερα το 14-6 που προβλέπει μέχρι το 2020 να καταργηθούν όσες επιδοτήσεις βλάπτουν το περιβάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις απρόβλεπτες επιπτώσεις κάποιων επιδοτήσεων. Αυτοί οι στόχοι, αυτές οι προθεσμίες έχουν ήδη καθοριστεί και εντός της Ένωσης και διεθνώς Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να γίνουν σεβαστά. Τέλος. Διαφάνεια. Κύριε Υπουργέ, έχετε δυνατότητα να ανοίξετε τις πόρτες κάποιων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών. Τι θα κάνετε για τους πολίτες της Ένωσης. Πώς θα τους επιτρέψετε να ενημερώνονται να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις διαδικασίες και διαπραγματεύσεις για να μπορέσουν και αυτοί να συμβάλλουν σε αυτές. Ευχαριστώ πολύ.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 Τέσσερι ολόκληρε ερωτήσει. Εν πάση περιπτώσει, για το τελευταίο σημείο για τη διαφάνεια και το ανοιχτό πνεύμα, το πλούστερο είναι να κάνετε μια δήλωση ότι η Φιλανδική Προεδρία είναι προσιλωμένη στο ανοιχτό πνεύμα και εξασφαλίζουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση θα, είναι, ε, θα αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο και όλοι θα παρακολουθούμε τι διαπραγματεύσει. Αυτό είναι το πιο καλό. Ilmastonmuutos ihan, ε, ihan... Ναι. Πρώτα απ' όλα κλιματικές αλλαγές. Το χαρτοφυλάκιό μου ως Υπουργού και ως, ε, στη διάρκεια της ε, Φιλανδικής Προεδρίας είναι Γεωργία, Δάση, που είναι και το χαρτοφυλάκι όμω στην Φιλανδία και αλληλεία και άλλοι φυσικοί πόροι. Αυτές είναι λύσεις για τα πολέμηση των κλιματικών αλλαγών και των ε, προβλημάτων που έχουμε λόγω αυτών. Βιώσιμη χρήση των λευτικών πόρων μαζί με τις νέες τεχνολογίες ε, μας εξασφαλίζουν ε, μαζί και με την κυκλική οικονομία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και έτσι όλο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό το σύνολο όλων αυτών των τομέων ώστε να μπορέσουμε ε, να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις και πρέπει να τονίσουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα. Ήδη μίλησα για το EMFF, το σύστημα επιδοτήσεων που κάποιος το ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιδοτήσεις που να ε, διευκολύνουν την παράνομη ε, αλληλεία. Μπορεί κανείς ωστόσο να διαπράξει διάφορες παράνομες ε, πράξεις και γι' αυτό εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εκρίζωση των παρανομιών αυτών. Είναι και θέμα δικαιοσύνης, γιατί οι περισσότεροι φορείς λειτουργούν με βάση τη νομοθεσία. Ε, ε, θα ήταν άδικο το να μην διωχθούν οι παραβάτες. Οι λεπτομέρειες που αναφέρατε θα μας απασχολήσουν σίγουρα αργότερα και ε, ελπίζω ότι αυτό θα γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε και εδώ βεβαίως θα θέλαμε να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους για συνεργασία. Η Φιλανδία φυσικά κάνει κάθε προετοιμασία για όλα αυτά. και ε, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι από εδώ και στο εξής όσο γίνεται πιο ανοιχτή. Μια μικρή προσθήκη τώρα για τα ΤΑΚ. Ήδη το είπα, αλλά μπορώ να το επαναλάβω. να έχουμε δηλαδή συνεργασία για την κοινή αλληλευτική πολιτική χρειάζεται συνεπώς να χρησιμοποιούμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, επιστημονικά στοιχεία και αυτό αποτελεί εγγύηση όσον αφορά την προστασία των αλληλευτικών αποθεμάτων και το περιβάλλον αλλά και τους καταναλωτές. Είμαι λοιπόν ε, δεσμευμένος και προσιλωμένος στους στόχους μέγιστον βιώσιμων αποδόσεων. Δεν άκουσα όμως ε, τη δέσμευσή σας να ανοίξετε το συζήτηση για τα ΤΑΚ σε δημόσια ακρόαση. Έχετε όμως τρεις μήνες μπροστά σας μέχρι τότε. Ε, ελπίζω να μας εκπλήξετε ευχάριστα. Δύο ακόμα συντονιστές και μετά Έξι ε, μέλη ε, έχουν ζητήσει το λόγο. Θα κλείσω τον κατάλογο και μετά τους συντονιστές θα πρέπει να ομαδοποιήσω ε, τις ερωτήσεις για λόγο περιορισμού χρόνου. Παρακαλώ, κυρία Κόντε. Οι δικέ μου ερωτήσει θα είναι πολύ πιο απλέ. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον Υπουργό για το σημερινό διάλογο. Η Προεδρία θα πρέπει να ασχοληθεί με δύο θέματα πολύ σημαντικά. Ε, αναφέρομαι στην μέγιστη απόδοση και στον κανονισμό για, την, ε, για τους ελέγχους. Ε, Επίση, στο πνεύμα τη συνεργασία, στο οποίο αναφερθήκατε και εσεί προηγουμένω, θέλω να ρωτήσω αν έχετε σκοπό να δώσετε περισσότερο φωνή στον αλευτικό τομέα και να μην περιοριστείτε στην λήψη των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η εφαρμογή τη κοινή αλευτική πολιτική δίνει καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη Βόρεια Θάλασσα, χάρη στα ε, μέτρα τα οποία έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η αλληλεία στην Μεσόγειο αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες ε, σε όλους τους τομείς και θυμίζω ότι είναι τελείως διαφορετική από αυτήν της Βόρειας Θάλασσας. Πρέπει λοιπόν να προσεγγιστεί με, την, ε, με, τρόπο λόγω της ιδιαιτερότητάς της που συχνά ε, είναι αλληλεία μικρής κλίμακας. Πολύ συχνά οι αλληλείς ε, χρειάζεται να περιμένουν ε, και να τηρούν διατάξεις που είναι επιβαρυντικές. Αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα ανεργίας, κυρίως για τους νέους. Δεν μπορούμε δηλαδή να ξεχνάμε την κοινωνικο-οικονομική σημασία των μέτρων που λαμβάνονται. Θα πρέπει πάντοτε στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας ε, να είμαστε προσιλωμένοι. Το περιβάλλον αλλά και η ε, κοινωνία και η οικονομία. Ευχαριστώ. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kysymyksistä. Tämä laajalainen vuoropuhelu on, on ilman muuta se, se, mitä... Μάλιστα, σα ευχαριστώ. Ο ευρύς και βαθύς διάλογος μεταξύ θεσμών είναι αυτός που θέλω να τονίσω όσον αφορά την προετοιμασία της κοινή αλευτικής πολιτικής. Βεβαίως, τα κράτη-μέλη συζητούν ε, τι ε, πρέπει ε, να γίνει, αλλά και η Κομισιόν. Τα τρία κριτήρια της βιωσιμότητας θα πρέπει να εξετάζονται πάντοτε από κοινού, γιατί συνδυάζονται και αποτελούν την βιωσιμότητα αυτή καθ' αυτή. Δεν μπορούμε να εξετάζουμε έναν από αυτούς τους παράγοντες ξεχωριστά. Θα πρέπει ταυτόχρονα να τους εξετάζουμε όλους. Επίσης, έχω συχνά παρατηρήσει ότι ιδιαίτερα η δημόσια συζήτηση εξετάζει μία πτυχή βιωσιμότητας μόνο και έτσι ε, έχει μια στρεβλωμένη εικόνα της κατάστασης. Δεν έχει μια συνολική εικόνα μόνο αν δει κανεί και τα τρία κριτήρια της βιωσιμότητας, η οικολογία, η οικονομία και η κοινωνία, μπορεί να ε, δει στο σύνολο την βιωσιμότητα. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε ξανά και ξανά. Αυτή είναι η πυλώνες της βιωσιμότητας και αυτό είναι η βάση για τα όσα κάνει η Φιλανδία. Κυρία Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ. Αφού μιλήσουμε και για την ε, Δυτική Μεσόγειο και για τα στόκ, θα ήθελα να ξέρω εάν θα ξεκινήσει και συγκεκριμένο πλάνο για την Αδριατική. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά νομίζω, όπως είπατε, ότι στη διάρκεια της Προεδρίας σας θα αναλύσετε ακόμα μια φορά τις δυνατότητες αλίας στην Μεσόγειο. Αν λοιπόν πραγματικά το είπατε. Τι σκοπεύετε ακριβώς να κάνετε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. So, as Υπουργέ, όπως όλοι γνωρίζουμε, το θέμα της αντιρρητικής ε, έχει κολλήσει νομίζω στο Συμβούλιο. Εσείς περιμένετε να απελευθερωθεί ή θα προσπαθήσετε να το ξεπαγώσετε το θέμα ή θα περιμένει μέχρι την επόμενη Προεδρία.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 Όσον αφορά την Αντιρρετική, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλες πληροφορίες να σας δώσω. Όμως όσον αφορά την Δυτική Μεσόγειο, εκεί προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Και βέβαια προσπαθούμε να βρούμε λύση, όπως σας είπα, για να πετύχουμε τους ε, στόχους μας. Um, So do you think the Council will discuss the age? Πιστεύετε λοιπόν πως το Συμβούλιο θα συζητήσει το φάκελο της αδιατικής μέχρι τα Χριστούγεννα. Από ό,τι κατάλαβα, όχι. Puheenjohtaja, niin kuin sanottu, niin se asia on, se asia on jumissa tällä hetkellä ja en osaa tuohon vastata. Että... Δεν μπορώ να σας δώσω πιο συγκεκριμένη απάντηση για το ναι ή όχι. Ως Φιλανδός μπορώ να σας πω ότι θα το δούμε. Μάλιστα, κύριε Τόμασιτς, επειδή εγώ προέρχομαι από την Κροατία, φυσικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Αδιατική θάλασσα, αλλά απλά είμαι περίεργη. Η Αδιατική θάλασσα είναι πολύ μικρή και αυτό σας δημιουργεί πολλά προβλήματα. Για ποιο λόγο? Μάλλον γιατί είναι μακριά από τη Φιλανδία, λέει ο πρόεδρος. Πολύ καλή ερώτησή σας, αλλά δεν ξέρω αν ο Υπουργός θα μπορεί να το απαντήσει αυτό. Θέλετε να προσπαθήσετε ή μήπως όχι niin kaikkiin kysymyksiin pitää puheenjohtaja yrittää aina vastata sen asian osalta ja Ναι, βεβαίω πρέπει να προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, έχω να πω το ίδιο όπως και πριν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μελετήσουμε εις βάθος. Ε, η υπόθεση αυτή είναι, όπως είπαμε, παγωμένη. Και ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση να δούμε πώς μπορούμε μια συμβιβαστική. Βαντάλεν τώρα, ένα λεπτό. Ja, welkom eh, meneer de minister. Ik heb een vraag en ik heb een, eh, een oproep. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Εσείς, ε, θέλω να σας θέσω μια ερώτηση και να σας κάνω και μια έκκληση. Συμμερίζομαι τη βούλησή σας ε, να τοποθετήσετε τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο. Σύμφωνο, αλλά διαπιστώνω και ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν προγράμματα που αφορούν τα κοινοτικά έχουν όμως ε, ε, εγκαταστάσεις για ε, πάρκα αιωλικής ενέργειας. Πώς εσείς το βλέπετε αυτό από την πλευρά της αλληλείας, ποιες είναι οι επιπτώσεις ας πούμε στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τι γίνεται με τον ανεφοδιασμό σε ψάρια και εδώ ε, εγώ μιλώ για τη φωνή των αλλιών. Ε, πριν να εγκατασταθούν τέτοια αιωλικά πάρκα, είναι σωστό να αναρωτηθούμε για τις επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στον κόσμο της αλλίας. Και πιστεύω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα μιλήσουν για το ίδιο θέμα. Κάτι ακόμα το οποίο αφορά το Brexit που ελπίζω να μην γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει αν φτάσουμε σε Brexit άνευ συμφωνίας, έχετε το σκοπό να προστατεύσετε τα συμφέροντα των αλλιέων και να μην τα παραμελήσετε. Energy industry versus fishing industry and uh... Βιομηχανία της ενέργειας εναντίον της λευτικής βιομηχανίας. Τι γίνεται εάν γίνει Brexit άνευ συμφωνίας. Κυρία Σλάιερ Πιέρεκ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για τις κάτω χώρες αυτό που έθεσε και ο συνάδελφος. Δεύτερη ε, ερώτηση. χθε ακούσαμε πως τέσσερα μεγάλα ε, ρωσικά σκάφη αλλιεύουν στα ύδατά μας υπό παράνομη σημαία. Το γνωρίζετε αυτό. και σίγουρα δεν έφτασαν εν μία νυχτή. Μιλάμε για βιώσιμη αλληλεία, αλλά αυτό εσείς ξέρατε ότι έχει συμβεί. Ίσως θα μπορούσατε να δώσετε μια, ένα σαφές μήνυμα, να δωσετε ενα σαφες μηνυμα να εξηγησετε στους Ρώσους ότι έχουν μπει, έχουν, χρησιμοποιούν ε, σημαίες άλλων χωρών και αλλιεύουν με αυτές τις σημαίες. Ε, να τους εξηγήσετε τι σημαίνει δίκαιη αλληλεία. Ε, χρειάζεται επίσης εναρμονισμένη ε, αλληλεία, αλλά και αυτή η υπόθεση με τη Ρωσία πρέπει να ξεκαθαριστεί οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που το αναφέρατε. Γκοζάλες Κασάρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχετε θάρρος. Είστε και υπουργό Γεωργίας και Στα πλαίσια της Προεδρίας σας είστε υπέρ Δεν είναι όμως απόλυτα σαφές ποιες είναι οι πολιτικές ε, τις οποίες υποστηρίζετε για την ηλικία. Και άλλοι συνάδελφοι μίλησαν για το Ταμείο Αλίας εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για τις συμφωνίες που είναι ακόμη εκκρεμίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικές για την κοινωνική βιωσιμότητα του αλλαυτικών μας στόλων. Κυρίως εγώ μιλώ για τον στόλο της Γαλλικίας που έχει συμφωνήσει τη Γουινέα Μπισάου με την Μαυριτανία. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μαυριτανία που δεν επιτρέπουν την εκφόρτωση οπλιστές μας υφίστανται μεγάλες ζημίες. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω για τη συμφωνία με το Μαρόκο, διότι πρέπει να πω ότι με εξεπλάγει, διότι υπάρχει ένα σημείο συμφωνία αυτή που δεν το περιμέναμε. Διότι στις διάφορες συμφωνίες δεν περιλαμβάνεται η ελίψη του Μαρλούκου. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Εάν έχουμε συμφωνίες συμφωνίες, συνεργασίες και βιωσιμότητε με τρίτε χώρες δεν θα πρέπει εκ μέρους τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέπουμε να αλλάζουν μονομερώς κάποιοι όροι της συμφωνίας. Γι' αυτό επιτρέψτε μου ε, να σας ζητήσω να δείξετε θάρρος για να διορθώσετε ότι είναι κακό κείμενο σε τέτοιου είδους συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ. Μιλήσατε εδώ επανελειμμένα για βιωσιμότητα, οικολογία, ε, περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία. Όμως όταν τα θέματα ε, βιωσιμότητας της οικονομικής και της κοινωνικής ε, μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή γιατί στην περιφέρεια που προέρχομαι από τη Σικελία πολλές φορές έχει προαγηθεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα εις βάρος της οικονομικής και της κοινωνικής και γι' αυτό εύχομαι όντως να δοθεί μεγαλύτερο βάρος ε, στην οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα ε, να πω τώρα τα εξή ε, σε σχέση κυρίως με τον κανονισμό περί ελέγχων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στην πρώτη ανάγνωση είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της Προεδρίας εάν εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει να απλοποιηθεί το σύστημα ελέγχου στον τομέα αλίας χωρίς επιπλέον φόρτο διοικητικό και χωρίς ε, αμφισβητήσιμες διατάξεις όπως ας πούμε εισαγωγή ε, κάμερα ε, με κλειστό κύκλωμα, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό για τους αλληλείς και κυρίως έχει εφέ στην ιδιωτική ζωή των εργαζομένων. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω αν έχουν προβλεφθεί οικονομικά μέτρα για τη στήριξη την διάλυση ε, αλευτικών σκαφών, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αύξηση της αλληλευτικής προσπάθειας, αλλά και το να δοθεί ε, δυνατότητα στους αλληλείς να εργάζονται ε, σε υγιές εργασιακό περιβάλλον. Ευχαριστώ. το Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να επανέλθω στις παρατηρήσεις που έκανε η συνάδελφη και συγκεκριμένη κυρία Κόντε. Θα μιλήσω για την μικρή κλίμαξη παράκτια αλία. Στην ε, Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές που παραγνωρίζεται εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτικών και αυτή πλή... φύγει κατά πρώτο λόγο η παράνομη αλληλεία. Θα ήθελα να επανέλθω στο παράδειγμα του Ζεύτα. Θα έπρεπε πριν να υπογράψουμε τις συμφωνίες που έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να θέσουμε ως προηγούμενο τη διασφάλιση των ελευτικών πόρων της Μεσογείου. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως αναφορά την απασχόληση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ποιες είναι οι δεσμεύσεις που θα λάβετε για να μπορέσετε να αποκαταστήσετε την οικονομική ισορροπία και την οικολογητή αυτή τη δραστηριότητα τη αλληλείας μικρής κλίμακας. Ευχαριστώ. And Mr. Bartolo. Ο κύριος Μπαρτόλο. Ε, καλημέρα σε όλους. Ε, κύριε Υπουργέ, καταρχάς σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην ε, Επιτροπή Αλλιές για να συζητήσουμε για τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας και για τις προκλήσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο εξάμεινο. Εγώ προέρχομαι από την αντίθετη όχθη της Ευρώπης, από τη Λαμπεντούσα, που είναι ένα μικρό νησάκι ανοιχτά της Σικελίας. Γεωγραφικά η Σικελία έχει 260.000 χιλιόμετρα ακτές ε, και ο τομέας Αλλιές απασχολεί 8.000 κόσμο ε, που οδηγούν σε κύκλο εργασιών πάνω από 300 εκατομμύρια ο Σικελικός στόλος με χιλιάδες σκάφη στη διάθεσή του έχει συνήθως μικρές, μικρής κλίμακας ασκή και αυτό σημαίνει έναν παράγοντα στήριξης οικονομικό αλλά είναι και ένα χαρακτηριστικό ιστορικό ε, της Σικελίας μας. Αυτός ο τομέας όμως τα τελευταία χρόνια έχει ιδιαίτερα επιβαρυνθεί και ε, να σας πω την εμπειρία του συστήματος ΣΤΑΚ, ένα σύστημα το οποίο οφείλεται στην ε, αλληλεία στον Ατλαντικό και στον Τόνο. Δεν ε, μπορεί να αυτό το σύστημα να εφαρμοστεί στην Μεσόγειο, ιδιαίτερα στην Σικελία και στην Ιταλία, όπου γίνεται μικρής κλίμακας αλληλείας κυρίως, όπου ε, επίσης εξαρτώμαστε από την εποχικότητα του αλλιεύματος. Θα πρέπει να υπάρχει δε μία διαμεσογειακή συνεργασία. Η μείωση του στόλου ε, του αλευτικού στόλου της Ευρώπης απέναντι στον Αφρικανικό στόλο έχει, δηλαδή το στόλο των χωρών της Βόρειας Αφρικής έχει οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια της ε, θαλάσσιας πανίδας. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των ε, αλλιευτικών ε, πόρων για να μπορέσουμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα και βιώσιμα αποτελέσματα και διαρκή αποτελέσματα όσον αφορά τα αποθέματα. Είναι απαραίτητη η συνεργασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο και την διάσκεψη για τις θαλάσσιες περιφερειακές περιοχές μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για τις παράκτες περιοχές περιοχές. Πρόεδρος, μπορείτε να ολοκληρώσετε και να κάνετε την ερώτησή σας. Η ερώτησή μου είναι ότι ελπίζω πως θα υπάρξει μια στεναρή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με τη Φιλανδική Προεδρία, με τρόπο ώστε να ευνοηθούν οι μικρές, μικρής κλίμακας ε, ε, αλλιευτικές δραστηριότητες, αλλά και κυρίως για τις χώρες που λειτουργούν στη Μεσόγειο και που συνορεύουν με τις αφρικανικές χώρες. Well, No shortage of questions. ερωτήσεις έχετε. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και ειδικέ που μου θέσατε. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να απαντήσω. Θα αρχίσω από το θέμα των πηγών ενέργειας. Θέλουμε τις, ε, τα ορικά καύσιμα να μπορέσουμε να σταματήσουμε να το χρησιμοποιούμε. Θέλουμε εναλλακτικέ πηγές ενέργειας που δεν δημιουργούν τα τελευταία θερμοκηπίου. Θα πρέπει όμως να κάνουμε, να δούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις αλληλευτικές δραστηριότητες. Βρεθούν λύσεις και ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, αυτό είναι σαφές, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλες αξιολογήσεις. Τώρα, το θέμα του Brexit. Χθες το βράδυ ακούσαμε κάποια νέα Όλε οι εναλλακτικέ λύσει είναι ανοιχτέ. Δεν μπορεί να πει η Προεδρία τι θα συμβεί στο μέλλον. Οι αποφάσει για το Brexit λαμβάνονται σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και βεβαίω, αυτή τη στιγμή αναμένουμε την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Φινλανδία το γεγονός ότι αν συμβεί το Brexit θα έχει πραγματικές επιπτώσεις και στον τομέα της αλληλείας και στις ποσοστώσεις και στο ΤΑΚ για όλους και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά η αλληλεία είναι μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που θα επηρεαστεί στα πλαίσια του Brexit. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες σενάρια όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναλύουμε τα διάφορα θέματα, αρμοδιότητες μας, από κοινού με τα άλλα κοινοτικά όργανα. Αυτό μπορώ να πω προς το πάνω. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Αλλά, επαναλαμβάνω, είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εναλλακτική λύση. Επόμενη ερώτηση. Οι παράνομες αλληλευτικές δραστηριότητες της Ρωσίας. Όποιος και να κάνει τέτοιου είδους δραστηριότητες θα πρέπει να ξέρει ότι μόλις ανακαλυφθεί τι κάνει θα γίνει κάτι διότι αυτού τέτοιου είδους πρακτικές είναι παράδεκτες. Τώρα, συμφωνίες με τρίτες χώρες. Συνεχίζουμε να παρατείνουμε τέτοιου είδους συμφωνίες, να τις ανανεώνουμε. Τα προβλήματα με την ε, συμφωνία με το Μαροκό δεν τα γνωρίζουμε. Καλό είναι να γίνει και εδώ διάλογος, αλλά ο κύριος κανόνας ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να παρατείνουμε τέτοιου είδους συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Η απλοποίηση. Όσον αφορά τον κανονισμό ελέγχου της Αλίας, όντως θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά, αποδοτικά μέτρα. Αυτό είναι μέρος του επόμενου PDP και υποστηρίζουμε τα λευτικά σκάφη και τους ελέγχους. Επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της σωστής λήψης και τη εισοδημάτων των ελιαίων όλο και περισσότερο γυράσκουν οι αλείς, όλο και λιγότερους νέους αλείς έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε και εδώ την κατάλληλη ισορροπία. Τώρα όσον αφορά την ε, μικρές κλίμακας αλίευση. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Επίσης, η διασυνοριακή συνεργασία στην Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές όπου γειτονεύουμε με τρίτες χώρες είναι κάτι που μας απασχολεί. Στην ε, Φιλανδία το γνωρίζουμε το πρόβλημα με τη Βόρεια Θάλασσα και με γείτονες τρίτων χωρών. Και βεβαίως πρέπει πάντα να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις ώστε να είναι εποφελείς οι δραστηριότητες, οι αλληλευτικές τους τρεις τομείς που προανέφερα. Σας ευχαριστώ. Καλύψατε πολλά θέματα σε μικρό χρονικό διάστημα, κύριε Υπουργέ. Θέλει κανείς να επανέλθει σε κάποιο θέμα. Ναι, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, λέει η κυρία ε, θα σας δώσω λεπτομέρειες όσον αφορά αυτά τα λιευτικά σκάφη, ε, ρωσικά. Βλέπω ότι εσείς είστε υπουργό Γεωργίας, Οκομίας και Αλίας. Εμείς ε, έχουμε κάπως διαφορετική κατάσταση στην ε, Ολλανδία. Εσείς μιλάτε για την κλιματική αλλαγή. Στο άρθρο 2 αναφέρεται επίσης και η ασφάλεια των ε, ειδών διατροφής και πάντα γίνεται λόγος για την αλληλεία, για τους αλλιευτικούς πόρους. Η ασφάλεια των ειδών ε, διατροφής επίσης είναι πρωταρχική σημασία και τα αλλιεύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των ειδών διατροφής. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στο γεγονός ότι θα πρέπει τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα να επιμείνουν σε αυτά τα θέματα. Είμαι υπέρ της προστασίας του κλίματος αλλά δεν έχουμε επαρκή παραγωγή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς πρέπει να προστρέχουμε σε αλλιεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό ήθελα να πω. Okay. Point, point, point made, I think. Uh, Ωραία παρατήρηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις εγώ. Πρώτα απ' όλα, αναλάβατε στην αρχή της συνεδρίας προσωπικές δεσμεύσεις για τα τάξ και για το... Ε, περίφημη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κοντά στο στόχο. Τον Δεκέμβριο στην συνεδρίασή μας θα έχουμε τελευταία ευκαιρία, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε του χρόνου να ολοκληρώσουμε αυτές τις προσπάθειες. Εσείς προσωπικά θα πρέπει να επιμείνετε ώστε να ακολουθούν οι, τα κράτη-μέλη τις επιστημονικές, τα επιστημονικά αποτελέσματα και ευρήματα. Δεύτερον, Νομίζω ότι θέλουμε άνοιγμα στον τρόπο με τον οποίο ληφθούν αποφάσεις και το Δεκέμβριο. Λέγει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτέ οι συνεδριάσει των ε, Υπουργών όταν νομοθετούν. Ίσως δεν πρόκειται για, να, για νομοθετικές πράξεις, ε, παρόλο που περί αυτού πρόκειται ακόμη όταν συζητείτε διάφορους κανονισμού. Λοιπόν, άνοιγμα, άνοιγμα. Μπορείτε τέτοιου δεσμεύσεις να τις αναλάβετε. Όταν υποβάλλετε προτάσεις και συζητήσεις θα μπορούσατε ανοιχτά να συζητείτε, συζητάτε συγγνώμη, για κάποια θέματα ε, πριν να λαμβάνετε τις αποφάσεις σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πρόσθετες ερωτήσεις. Είναι σαφέ σαφές ότι κανένας δεν θα πρέπει να ξεφεύγει χωρίς κυρώσεις όταν κάνει, έχει μια δραστηριότητα παράνομη. Η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η αλληλεία είναι μέρος όλου του συστήματος παραγωγής ειδών διατροφής με ασφάλεια για τους καταναλωτές. Επίσης ο πρόεδρος μίλησε για επιστημονικά ευρήματα και ενδείξεις. Είναι απόλυτα σαφές. Θα πρέπει να, για αυτά τα θέματα να ευρεθεί πολιτική συνένεση. Διαφορετικά ποτέ δεν θα μπορέσουμε για τις ποσοστώσεις και τα τάξη να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Η Φινλανδία τηρεί την αρχή αυτή και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να προχωρήσουμε. Βεβαίως, βάσει επιστημονικών δεδομένων και βρημάτων. Και στα πλαίσια της βιωσιμότητας. Εμείς είμαστε υπέρ της τη της ανοιχτής σεβόμεθα και την κατανομή των εξουσιών μεταξύ των τριών κοινοτικών οργάνων και σεβόμεθα και την συνθήκη. Στα μέτρα του δυνατού βεβαίως όλα αυτά, ώστε με μέτρο να είναι όλα καλά. Καλό, καλό πράγμα είναι αυτό που λέτε για τα πάντα. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας αφιερώσετε κύριε Υπουργέ. Καλή τύχη στους επόμενους 3,5 μήνες της Προεδρίας σας. Σας ευχαριστώ. Θα συνεδριάσουμε και πάλι στις 2,5 λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ συνάδελφοι.